Αρχίζουμε εκ νέου τη συνεδρίασή μας και θα ήθελα να αρχίσουμε με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η ψηφοφορία στον έλεγχο από τα κράτη-μέλη των εκτελεστικών εξουσιών της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να, ρωτήσω τον κύριο, να ζητήσω από τον κύριο Αλμπερτίνη να κάνει μια δήλωση θα ήθελα επίσης να επισύρω την προσοχή των συναδέλφων ότι αυτή δεν, είναι, δεν πρόκειται για συζήτηση. Πρέπει να ψηφίσουμε, άρα θα θέλαμε ο κύριος Αλμπερτίνη να κάνει τη δήλωση που επιθυμεί και αν υπάρχει παρέμβαση από τους συναδέλφους να είναι πολύ σύντομη γιατί πρέπει να ψηφίσουμε. Έχουμε μία κοινή συζήτηση, μία κρόαση στη συνέχεια και θα ήθελα τώρα ο κύριος Αλμπερτίνη να κάνει εν συντομία τη δήλωση που επιθυμεί. Ευχαριστώ. Δύο κουβέντες μόνο για να σας πω πώς έχει το εν λόγω θέμα. Όπως ξέρετε το άρθρο 291 των συνθήκων για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εισήχθη από τη συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα ελέγχου των εκτελεστικών πράξεων και εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό βεβαίως θα πρέπει να συνάδει με τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως συνομοθέτου. Άρα αυτές οι δύο απαιτήσει συμβαδίζουν και για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να ασκήσει τα προνόμια αυτά και σε σχέση και με την ενδεχόμενη προσφυγή στο ΔΕΚ επί του θέματος, δηλαδή ως προς τα εκτελεστικά, τις εκτελεστικές εξουσίες, θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει επίσημα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάθε ενδεχόμενο μέτρο που προτίθεται να λάβει δυνάμει του άρθρου 291. Αυτή η διαδικασία πληροφόρησης είναι συμπληρωματική με αυτήν που προβλέπεται στον τρόπο λειτουργίας της ε, επιτροπολογίας. Δεν γίνονται διακρίσεις μεταξύ κατεξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων ή πράξεων εκτέλεσης και θεωρούμε ότι η γνωμοδότηση αυτή που θα ψηφιστεί σήμερα καθότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θα ψηφίσει αύριο άρα θα πρέπει εμείς να γνωμοδοτήσουμε ως λίμπε καταρχήν θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιβεβαιώσει τα προνόμια του ως συνομοθέτου δυνάμει του άρθρου 291 της Νέας Συνθήκης ως προς την αρμοδιότητα των κρατών μελών για την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ναι, έχετε το λόγο. Κύριε Λόισινγκ, η ομάδα μου θα υπερψηφίσει την έκθεση. Ωστόσο, θα προτιμούσαμε πολλά πράγματα που έχουν σχέση με τον εκδημοκρατισμό να είχαν διατυπωθεί με σαφέστερο τρόπο. Εκπλήσωμε για το γεγονός ότι όλες οι τροπολογίες των πράσινων προτείνεται να καταψηφιστούν από τον εισηγητή. Και τροπολογίες, μάλιστα, οι οποίες αρχικά είχαν προταθεί από τους φιλελεύθερους ή από τους χριστιανοδημοκράτες, αρχικά είχαν εγκριθεί από τον εισηγητή, τώρα που επαναφέρονται με παρόμοιο περιεχόμενο από τους πρασίνους, απορρίπτονται από τον ίδιο. Κάποιο πρόβλημα όμως φάνηκε να υπάρχει με την Ιταλική διερμηνία. Είναι εντάξει τώρα. And we'll start... Ο Προεδρεύων θα αρχίσουμε. Μα το είχα ανοίξει. Σας πιστεύω, εσείς τα βλέπετε καλύτερα το φωτάκι. Αρχίζουμε λοιπόν με την τροπολογία 17. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Σας ευχαριστώ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται 20 υπέρ κατά ευχαριστώ απορρίπτεται 21 ε, υπέρ κατά απορρίπτεται οι πέντε τώρα οι πέντε. υπέρ κατά εγκρίνεται υπαριθμών 6 υπέρ κατά εγκρίνεται υπαριθμών 7 υπέρ κατά εγκρίνεται 22 υπέρ κατά νομίζω ότι χρειάζεται επαλήθευση παρακαλώ ηλεκτρονική, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 22 Βάλτε παρακαλώ τις κάρτες σας. Έχει καλός. Τώρα λίγη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε. 23 αρχίζει η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πέρας. Απορρίφθηκε. 24 υπέρ. Κατά. Χρειάζεται και εδώ επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται αυτή. Υπάρχει μόνο 8 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται αυτή. 26 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά απορρίπτεται 10 υπέρ κατά απορρίπτεται και αυτή Ίσως είναι δυνατόν να ψηφίσουμε την 11, 12 και 14 μαζί, αν συμφωνείτε. Υπέρ της 11, 12 και 14 κατά. Απορρίπτονται και οι τρεις αυτές τροπολογίες. 13. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη 1. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά εγκρίνεται αυτή 16 υπέρ κατά απορρίπτεται 2 υπέρ κατά εγκρίνεται 3 υπέρ κατά εγκρίνεται 4 υπέρ κατά εγκρίνεται 9 υπέρ κατά απορρίπτεται η τελική ψηφοφορία επί του σχεδίου γνωμοδοτήσεως όπως ο πήθηκε ονομαστική ηλεκτρονικά επομένως αρχίζει πέρας ε, εγκρίνεται λοιπόν και συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία πρόταση εκ μέρους σοσιαλιστών και δημοκρατών. Αύριο υποτίθεται ότι ψηφίζουμε Αύριο υποτίθεται ότι ψηφίζουμε το ψήφισμα για την ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Αλβανίας. Γνωρίζετε ότι τις τελευταίες εβδομάδες οι δύο ηγέτες των ε, κομμάτων των βασικών της Αλβανίας, CPP και SMD, προσπαθούν να φτάσουν σε κάποιο συμβιβασμό, αλλά δυστυχώς δεν τα έχουν καταφέρει ακόμη. Από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Ντόλ πρόκειται να πάει στην Αλβαλία και να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και άλλους ηγέτες. Θεωρώ ότι αν θα αναβάλουμε την ψηφοφορία την αυριανή, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τον κύριο Ντόλ και το Κοινοβούλιο στο να βοηθήσουν στην επίτευξη μιας ε, κοινή λύση για την Αλβανία. Νομίζω ότι δεν θα στείλουμε το κατάλληλο μήνυμα αν συνεχίσουμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Γι' αυτό προτείνω αναβολή της ψηφοφορίας για τον Ιούλιο και ελπίζουμε ότι μέχρι τότε θα έχουμε καταλήξει σε συμβιβασμό. Ευχαριστώ. Η κυρία Πακ. Συζητήσαμε ήδη το αίτημα αυτό των σοσιαλιστών. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αναβάλουμε για δεύτερη φορά έκθεση περί Αλβανίας για τον Ιούλιο. Δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει εκλεγμένη κυβέρνηση στην Αλβανία, υπάρχει Βουλή, όπου πηγαίνουν ξανά οι σοσιαλιστές, έχουν ξαναλα... ξανακαταλάβει τις θέσεις τους εκεί, λειτουργεί η Αλβανική Βουλή. Τα προβλήματα δεν εντοπίζονται στο Κοινοβούλιο εκεί, αλλά σε εντελώ διαφορετικό χώρο. Όσοι ασχολούνται με το θέμα γνωρίζουν καλά τι συμβαίνει. Αυτά που αναμένουμε από την κυβέρνηση είναι να πράξει μαζί με την αντιπολίτευση αυτά που συζητήθηκαν ήδη μεταξύ Ντόλ και Σούλτς. Δηλαδή να μελετήσει νέο εκλογικό νομοσχέδιο Υπάρχει εκλογικό νομοσχέδιο το οποίο έχει συζητηθεί ήδη από διετία. Φαίνεται πως δεν ικανοποιεί ωστόσο την αντιπολίτευση, γι' αυτό και η κυβέρνηση και το δεύτερο κόμμα που συναπαρτίζει την κυβέρνηση έχουν δηλώσει την διάθεσή τους για το μέλλον να συζητήσουν νέο εκλογικό νομοσχέδιο. Αλλά το παρελθόν είναι παρελθόν. Οι εκλογέ που έγιναν πέρσι θεωρήθηκαν, κρίθηκαν από όλου ω ορθέ, ω σωστέ. Όλοι οι εκλογικοί παρατηρητές ανεγνώρισαν τις εκλογές αυτές. Μόλις αργότερα αποφάσισε ο επικεφαλή της αντιπολίτευσης εκεί ότι έπρεπε να είχαν ανοίξει οι κάλπες. Το να ανοίξουν οι κάλπες δεν είναι υπόθεση της Βουλής. Είναι παράνομο. Είναι παράνομη πράξη. Και άλλωστε δεν το συζητούν πλέον καν αυτό οι αρχηγοί Ντόλ και Σούλτς. Αυτά που πρέπει να επιτευχθούν ή θα έπρεπε να επιτευχθούν μέσω των συζητήσεων αυτών θα είναι να επιστρέψουν στην Βουλή όλοι και να βάλουν στον δρόμο του το νομοσχέδιο. Ακόμα και αν αναβάλουμε εμεί την έκθεση, δεν επηρεάζουμε τη διαδικασία αυτή ούτε προ τη μία ούτε προ την άλλη κατεύθυνση. Το σωστό θα ήταν να ψηφιστεί αύριο η έκθεση Κάοπη και να συμβάλλουμε ώστε να ξεφύγει πλέον η χώρα από την κρίση. Προβλήματα θα έχει ίσως Πάντα υπάρχουν προβλήματα και σε άλλες χώρες που δεν είμαστε τόσο επικριτικοί απέναντί τους. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε να κάνουμε διάκριση για την Αλβανία και επομένως να μην είμαστε και δίκαιοι απέναντι σε μια εκλεγμένη κυβέρνηση και σε ένα εκλεγμένο κοινοβούλιο εκεί. Κύριε Νέιτς. Κύριε Πρόεδρε, σε αντίθεση με την κυρία Πακ, η πλειοψηφία στη δική μου πολιτική ομάδα, αν και όχι το σύνολο των συναδέλφων, θα ήθελε να δώσει μια τελευταία ευκαιρία, γι' αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε στην αναβολή. Ευχαριστώ η κυρία Νίλσεν. Ευχαριστώ. Εν συντομία, εμείς θα συμφωνήσουμε με την θέση του συγητή. Αν προτιμούν αναβολή, θα συμφωνήσουμε. Ο κύριος Πρέντα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Με τον συντονιστή τον κύριο Σαλαφράνκα αποφασίσαμε να συμφωνήσουμε με την κυρία Πακ αν και δεν θεωρούμε ότι υπάρχει σαφής δικαιολογία. Ο κύριος συζητητής, κύριος Χουντής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θυμίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι πριν από τρεις εβδομάδες υπήρξε κοινό αίτημα, επαναλαμβάνω κοινό αίτημα όλων μας, να υπάρξει αναβολή ούτω ώστε στο μεσοδιάστημα να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τώρα το αίτημα φαίνεται ότι δεν είναι κοινό. Και το λέω αυτό γιατί σε όλη την προσπάθεια και ευχαριστώ για άλλη μια φορά τους σκιώδεις συζητητές, στην έκθεση αποπειραθήκαμε και έχουμε κάνει καλή δουλειά όλοι μαζί και έτσι βοηθάει όλη αυτή την υπόθεση. Ε, η δική μου γνώμη είναι αφού δεν υπάρχει κοινό αίτημα δεν νομίζω πως είναι σωστή μια δεύτερη αναβολή. Μια δεύτερη αναβολή θα φέρει, δεν συνηθίζεται, δεύτερο θα φέρει πολύ πίσω την τελική ψήφιση με συνέπεια το Σεπτέμβριο να χρειαστεί μια καινούρια έκθεση που θα επικαιροποιήσει αρκετά από αυτά που σήμερα διατυπώνουμε κατά τον τρόπο που διατυπώνουμε. Δεν υποτιμώ καθόλου τις προσπάθειες που γίνονται και αυτό το διάστημα. Και επειδή από ό,τι είδα θα γίνουν επισκέψεις αυτή την εβδομάδα. Αν υπάρξουν αποτελέσματα πράγματι που το ευχόμαστε, όλοι, μπορούμε στην Ολομέλεια του Στρασβούργου με προφορική τροπολογία να αποτυπώσουμε τα θετικά αποτελέσματα που ενδεχομένως θα έχει, όπως επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, εύχομαι να έχει αυτή η επίσκεψη. Ε, επομένως η δική μου γνώμη είναι να μην αναβάλουμε για δεύτερη φορά την ψήφιση αυτής της έκθεσης και να προχωρήσουμε κανονικά. Ευχαριστώ. Καλά. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η ψηφοφορία θα γίνει αύριο κανονικά. Έχουμε το Λαϊκό Κόμμα, την Ενωτική Αριστερά και τους Πράσινους που είναι υπέρ της διεξαγωγής ψηφοφορίας αύριο που φτάνουμε στα 37 μέλη σύμφωνα με τον κατάλογο που έχουμε εδώ και έχουμε και την άλλη άποψη που τάσσεται υπέρ της αναβολής. Και έχουμε και τους φιλελευθέρους οι οποίοι και αυτοί τάσσονται υπέρ της αναβολής. Εσείς κύριε Τάνοκ, δεν είχα σκόπο να παρέμβω, αλλά η γνώμη της ομάδας μου αλλάζει και θα συμπαραταχθούμε με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Άρα λοιπόν η πλειοψηφία τάσεται υπέρ της διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Ξέρετε τι θα γίνει αύριο. Εκτός εάν, εκτός εάν αλλάξουν πάλι γνώμη οι πολιτικές ομάδες μέχρι αύριο το πρωί. Ελπίζω να μην προεδρεύω εγώ. Άρα δεν θα είναι τότε δικό μου το πρόβλημα. Άρα τώρα πρέπει να αρχίσει η δημόσια ακρόαση. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα προχωρήσουμε στο βασικό θέμα της ακρόασής μας σήμερα. Θα ήθελα να προσκαλέσω τους εμπειρογνώμονες να έρθουν να καθίσουν εδώ.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 subito, se non <clears throat> Αγαπητοί συνάδελφοι, με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα να ε, αρχίσω με αυτή την ακρόαση σε σχέση με την ε, Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική θεμάτων ασφαλείας. Ο κύριος Ντανζάν είναι συμπρόεδρος αυτής της ε, ακρόασης είναι η καταλληλότερη στιγμή για να μιλήσουμε για αυτή την πρωτοβουλία. Αρχίζουμε με ένα προηγμένο στάδιο σκέψεων για την μεταρρύθμιση των δύο αυτών βασικών οργανισμών, δηλαδή του ΝΑΤΟ και του ΟΑΣΕ. Αυτό είναι και ο στόχος αυτής της ακρόασης και υπάρχει και μια πρόταση ψηφίσματος για το τέλος των συζητήσεων. Τον Νοέμβριο οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων των χωρών ΝΑΤΟ θα συζητήσουν σε μια διάσκεψη κορυφή στη Λισαβόνα ε, θέματα εξέλιξης του ΝΑΤΟ. Στις 27 Ιανουαρίου το συζητήσαμε με την Ματλέν ε, Ολμπράιτ που είναι επικεφαλής των εμπειρογνωμόνων για το σενάριο αυτό μετεξέλιξης του ΝΑΤΟ. Ε, ως προς το Νοασέ, το Καζακστάν έχει την προεδρία, κατέχει την προεδρία και θα προετοιμάσει μία διάσκεψη κατά το τέλος του έτους. Άρα θα ήταν σκόπιμο να προωθήσουμε και εμείς τα δύο αυτά θέματα. Η τελευταία μεταρρύθμιση των δύο αυτών οργάνων έγινε το 1999. Στα 17 χρόνια έχουν επέλθει μεγάλες αλλαγές. Ε, γνωρίσαμε πολλές απειλές, τρομοκρατικές δραστηριότητες στο τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Η Ευρώπη άλλαξε μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και με την προσχώρηση νέων κρατών μελών, άρα θα ήταν σκόπιμο να μας απασχολήσει αυτό το ζήτημα και αυτή είναι η καταλληλότερη στιγμή. Θα μας απασχολήσει αυτή η παράλληλη διαδικασία μεταρρύθμισης, λαμβάνοντας υπόψη και την πρόταση Μετβέντεφ για μια Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ασφάλειας, για να εξετάσουμε κατά πόσο κινούμαστε σε μια νέα ευρωατλαντική δομή ασφάλειας. Θα ήθελα να αφήσω την απάντηση σε αυτό το ερώτημα στους συνομιλητές μας. Ο καθηγητής Σιλβέστρη που είναι πρόεδρος της Επιτροπής ε, της Ρώμης Διεθνών Μελετών ο, ο κύριος Νταν ε, Χάμιλτον του, από το John Hopkins και στην κυρία Μάρα Μαρινάκη της ε, μόνιμης αντιπροσωπείας, από τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΑΣΕ και την κυρία Αρμπατόβα η οποία ασχολείται με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Μελετών της Μόσχας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ε, συνομιλητές και θα αναθέσω την Προεδρία στον συνάδελφο Πασκού. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή εργασία. I would like to ask Mr. Θα παρακαλέσω τον κύριο Στέφανο Σιλβέστρη να λάβει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα τα πω λοιπόν λίγο συνοπτικά. Ναι, είναι αναποφευκτό άλλωστε αυτό. Διαγράφεται μια διαδικασία προσαρμογής στο νέο διεθνές σενάριο, αλλά δεν έχουμε φτάσει κατά τη γνώμη μου ακόμα στο σημείο αυτό. Βλέπουμε μια γενικευμένη κρίση των οργανώσεων ε, άμυνας και ασφάλειας που προσπαθούν να προσαρμοστούν στα σενάρια που αλλάζουν αλλά για δύο λόγους, αφενός γιατί είναι δύσκολη αλλαγή αυτή και διότι αφετέρου δεν είναι και σαφές, σαφής η αντίκτυπη των αλλαγών στις διάφορες ε, πραγματικότητες ε, γεγονός είναι εν πάση περιπτώσει ότι οι αλλαγές αυτές δεν φαίνονται ιδιαίτερα πιστικές. Εάν εξετάσετε την έκθεση των σοφών του ΝΑΤΟ, της Επιτροπής δηλαδή Όλμπραϊτ για την μεταρρύθμιση του ΝΑΤΟ, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις νέες απειλές. Η ανταπόκρισή τους είναι λίγο πολύ τα πάντα. Δηλαδή βάζουν κάτω ολόκληρο το μενού ή εν πάση περιπτώσει ένα μεγάλο μενού αν θέλετε, ένα μεγάλο κατάλογο όλων των πιθανών επιλογών. Δεν είναι βέβαια μόνο δικό τους το πρόβλημα. Αν δείτε και την ανατετραετία uh, Defense Review του Πενταγώνου κατά κάποιο τρόπο αν και κατά κάποιο τρόπο καλύτερα δομημένα τα λένε όμως τα ίδια πράγματα εν τέλει Κάποτε η ιδέα του Πενταγώνου ήταν η ικανότητα να διεξάγει ενάμιση πόλεμο ταυτόχρονα, ενάμιση με δύο. Τώρα προτείνουν τρία περίπλοκα σενάρια. Κάθε ένα από αυτό με διαφορετικές αναμίξεις πολεμικών μετόπων, με ταυτόχρονη ε, μείζωνα επιχείρηση σταθεροποίησης, η υποστήριξη ε, αμερικανικών μη στρατιωτικών αρχών ε, για την αντιμετώπιση θεομηνιών, ανθρωπιστικών ε, επιγουσών περιπτώσεων κτλ. Το δεύτερο, δύο περιφερειακά, μέτωπα συν μια σημαντική επιτήρηση μέσα και γύρω από τις ΗΠΑ και το τρίτο σενάριο μια μεγάλη σταθεροποιητική επιχείρηση μεγάλης διάρκειας συν αποτροπή σε ξεχωριστό θέατρο συν άλλες αποστολές μικρότερου ε, πιο περιορισμένου χαρακτήρα. Και εδώ λοιπόν πάλι η συνταγή είναι λίγο απ' όλα. Η ιδέα είναι ότι θα πρέπει να διατηρεί κανείς μια ευελιξία διότι ποτέ δεν ξέρεις. Ο αριθμός των πιθανών εχθρών είναι μεγάλος και ποικίλος. Οι περισσότερες νέες απειλές δεν είναι ξεκάθαρες γεωγραφικά. Είναι μεγάλο το πλήθος των πιθανών σεναρίων και μεγάλο το πλήθος των ε, πιθανών επιλογών. Για να θυμηθούμε τι έλεγε παλαιότερα ο Ράμσφελντ, δεν ξέρουμε ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Μέσα σε αυτή την κατάσταση είναι πολύ δύσκολο να γίνει ξεκάθαρο σχεδιασμό και ξεκάθαρη μεταρρύθμιση. Τι σημαίνουν αυτά. Σημαίνουν ότι η Ατλαντική Συμμαχία κάνει ταυτόχρονα και το στρατηγικό τη στόχο και το γεωγραφικό τη πεδίο ε, ανάπτυξης. Δηλαδή δεν έχει ούτε ξεκάθαρο εχθρό, ούτε δεν ξέρει πού θα κληθεί να δράσει. Το γεγονός ότι ο, μόνο, ο μόνος πόλεμος που διεξάγει μονο πόλεμο μονος που διεξαγει αυτη τη στιγμή είναι εκτός των ορίων της συνθήκης της Ουάσιγκτον είναι και μια ξεκάθαρη ένδειξη για αυτό που λέω. Τι σημαίνει αυτό τώρα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Δεν λέει καλά πράγματα, γιατί η ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα χρειάζεται να βασίζεται σε μια αποτελεσματική σχέση με τις Ενωμένες Πολιτείες, διότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν στη διάθεσή τους έναν αριθμό ικανοτήτων και και οι προπολογισμοί τους είναι περιορισμένοι και οι αρμοδιότητες είναι κατακαιρματισμένε εθνικά. Το θετικό είναι ότι η νέα Αμερικανική Εθνική Στρατηγική που ε, αναπτύσσει ο πρόεδρος Ομπάμα απαιτεί και να υπάρχουν σύμμαχοι οι οποίοι να ανταποκρίνονται. Βασίζεται δηλαδή σε αυτό και κατά πάσα πιθανότητα θα δεχθούν και κάποια αποτετήματα των συμμάχων. Το πρόβλημα είναι ποιοι είναι οι σύμμαχοι. Είναι μια παρουσία των συμμάχων οι σύμμαχοι δεν είναι πραγματικά παρόντες στην Αντιλαντική Συμμαχία, ούτε και θα είναι στην παρούσα κατάσταση. Εν τέλει, νομίζω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση μία απλή μικρή τροποποίηση των υφισταμένων οργανώσεων που ασχολούνται με την ε, ασφάλεια και την άμυνα δεν θα μας δώσει πολύ πιο ξεκάθαρη κατάσταση, ξεκάθαρη και ασφαλή κατάσταση. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί μάλλον να δεχθεί την ιδέα ότι θα χρειαστεί να εκπονήσει ένα, μια βαθύτερη και σημαντικότερη στρατηγική ασφαλείας που να βάζει στο κέντρο της τα ε, συμφέροντα ασφαλεία Σε αυτή την κατάσταση δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση καλά θα κάνει να, αναγνωρίζει, να αναγνωρίσει μάλλον ότι βρίσκεται σε μια περίπλοκη γειτονιά. Η στρατική που χρειάζεται είναι μάλλον περιφερειακή και λιγότερο παγκόσμια. Αλλά η περιφέρεια στην οποία βρίσκεται γεωγραφικά η Ευρώπη είναι από τις πιο ε, περίπλοκες αλλά και από τις πιο μπελαλίδικε εντό εισαγωγικών από τη Ρωσία μέχρι την Αφρική και βεβαίω τη Μεσόγειο. Οι εξαρτήσεις και το ευάλωτο της Ευρωπαϊκής Ένωση είναι σημαντικά. Ενέργεια λόγω τρομοκρατία, λόγω κλιματικότητα, μετανάστευση λόγω περιφερειακών πολέμων που έχουν σημαντικούς αντικτύπους στι ε, πολιτικές αυτέ, λόγω ε, παρουσίας όπλων μαζική καταστροφή λόγω της μείωσης του επίπεδου ασφαλείας των στρατηγικών γραμμών επικοινωνιών. Στην κατάσταση αυτή μέσα είναι δυνατό να διεξαχθεί νέος διάλογος με τις ΗΠΑ που μάλλον είναι το ουσιώδες στοιχείο για την επίλυση του προβλήματος. Δεν μπορώ να φανταστώ νέα αρχιτεκτονική που να βασίζεται σε διαφορετική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΑΣΕ και του ΝΑΤΟ, χωρίς πρώτα να καταλήξουμε σε μια νέα συμφωνία, σε μια νέα συνεννόηση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό μάλλον είναι και το μεγαλύτερο ερώτημα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ε, ε, στο μέλλον. Νομίζω ότι εξήλυσα και τα 10 λεπτά μου. Σας ευχαριστώ κύριε Σιλβέστρη θα παρακαλέσω τον κύριο Χάμιλτον να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς και τους συναδέλφους σας για την πρόσκλησή σας. Το θέμα μου είναι η αρχιτεκτονική της ασφαλείας. Οπότε θα ήθελα να σας μιλήσω για τους βασικούς πυλώνες της ΟΑΣΕ, ΝΑΤΟ, αλλά όπως είπε και ο Στέφανο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν ξεκινήσω να πω ότι υπάρχουν κάποια βασικά σημεία που θέτουν το πλαίσιο της συζήτησης. Καταρχάς, η Ευρώπη είναι πιο ολοκληρωμένη, πιο ελεύθερη και πιο ειρηνική από ό,τι εδώ και πολύ καιρό. Αλλά δεν είναι ούτε ολόκληρη, ούτε ελεύθερη, ούτε ειρηνική αν μιλήσουμε για το σύνολο του γεωγραφικού χώρου και υπάρχουν πολλές προκλήσεις εντός αυτού του γεωγραφικού χώρου αλλά και εκτός του που πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας. Τέλος, να πω ότι πιστεύω ότι πρέπει πάντα να, να θυμόμαστε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ευρωπαϊκή δύναμη. Και γι' αυτό το λόγο χαίρομαι ιδιαίτερα για την πρόσκλησή σας σε εμένα. Βλέποντας λοιπόν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, διαπιστώνουμε ότι οι θεσμοί μας και τα εργαλεία μας δεν είναι τα κατάλληλα. Έχουμε όμως την ιστορική ευκαιρία να καταφέρουμε κάτι, αλλά δεν το έχουμε κάνει ακόμη. Ξεκινάμε με τον πρώτο πυλώνα, τον ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι πιο πολυάσχολο από ποτέ. Αυτή τη στιγμή εμπλέκεται σε έξι αποστολές ταυτόχρονα, ενώ κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου δεν είχε ρίξει ούτε σφαίρα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι ακριβώς κάνει το ΝΑΤΟ. Όπως είπε και ο Στέφανο, υπάρχουν εκθέσεις και φαίνεται ότι μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να συνοψίσουμε, να απλοποιήσουμε το σκοπό του ΝΑΤΟ. Εγώ όμως νομίζω ότι είναι απλός αυτός ο σκοπός. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί στόχοι που παραμένουν από την ίδρυσή του. Τρεις κατά τη γνώμη μου πολύ απλοί. Καταρχάς, το ΝΑΤΟ είναι ο χώρος για τη συλλογική άμυνα των μελών του. Δεύτερον, ότι θεσμοποιεί τον διατλαντικό σύνδεσμο και δημιουργεί ένα φόρουμ για τη συνεργασία των εταίρων. Και τρίτον, κάτι που ξεχνάμε κατά καιρού στην ιστορία, είναι ότι παρέχει στους Ευρωπαίους διασφάλιση για τον εαυτό τους και για τις διαδράσεις μεταξύ τους τους ε, δίνει την εμπιστοσύνη που χρειάζονται για να μιλάτε για κοινή ασφάλεια χωρίς να φοβούνται ο ένας τον άλλον. Αυτό ήταν ένας από τους βασικούς στόχους του ΝΑΤΟ και ήταν και ένα μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ξεκίνημά της. Άρα, Τώρα το ΝΑΤΟ χρειάζεται νέες στρατηγικές έννοιες. Το καλύτερο είναι να συνοψίσουμε στα βασικά. Εγώ και οι συναδέλφοί μου πέρυσι παρουσιάσαμε μια έκθεση που προσπαθεί να κάνει αυτό ακριβώς και αναφέρει ότι ουσιαστικά το ΝΑΤΟ έχει δύο βασικά είδη αποστολών. Ορισμένες εκτός συνόρων, ορισμένες εντός του βορειοατλαντικού χώρου. Και πρέπει να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των δύο. Τα τελευταία 15 χρόνια δεν υπήρξε τόσο μεγάλη ισορροπία γιατί είχαμε περισσότερη έμφαση στα εξωτερικά. Όμως, αν σήμερα ρωτήσετε το κόσμο για τις ανασφάλειες τους εντός της χώρας του, εκεί το ΝΑΤΟ ακούγεται κάπως άσχετο. Χρειάζεται λοιπόν μια νέα ισορροπία εδώ. Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να ασχοληθεί πλέον και με θέματα όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η τρομοκρατία κτλ. που είναι σημαντικά, αν και εκεί ίσως το ΝΑΤΟ να μην παίξει τον κεντρικό ρόλο και επίσης την ειρήνη στην Ευρώπη είναι κάτι ακόμη όπου μπορεί να παίξει ρόλο το ΝΑΤΟ. Και εδώ πρέπει να θυμόμαστε ότι για να έχουμε μία ασφάλεια βορειοατλαντική, μόνο το ΝΑΤΟ είναι αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει. Αυτό πρέπει να παίξει τον ηγετικό ρόλο. Όμως, Σήμερα, όταν μιλάμε για εξωτερικές απειλές, δεν μιλάμε μόνο για στρατούς. Υπάρχουν και άλλες απειλές και γι' αυτό πρέπει το ΝΑΤΟ να μπορεί να συνεργαστεί και με πολλούς διαφορετικούς εταίρους. Είτε Ευρωπαίους, είτε Ρώσους, είτε και άλλους συμμάχους, όπως διαπιστώσαμε και στο Αφγανιστάν, οι οποίοι θα συνενώσουν τις, ομάδες, τις δυνάμεις τους μαζί μας. Κάτι που μέχρι σήμερα δεν το έκανε πολύ καλά το ΝΑΤΟ. Επίσης πρέπει το ΝΑΤΟ να είναι σε θέση να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση εκ των υστέρων σε συνεργασία με, τη, με τις πολιτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό πλαίσιο και πρέπει να δούμε και που έχει την ηγετική θέση το ΝΑΤΟ και που όχι. Κάτι άλλο που ανέφερε ο Στέφανο και θα ήθελα να αναφέρω και εγώ. Νομίζω ότι υπάρχει ρόλος για την σχέση ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει έναν τεράστιο χώρο όπου πολύ απλά δεν υπάρχουν πόλεμοι. Αυτή είναι πολύ βασική συνεισφορά. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι η βασική μας εταίρη. Ωστόσο δεν έχουμε στρατηγική σχέση. Είναι σημαντική η σχέση μας αλλά δεν είναι στρατηγική. Εξακολουθούμε να μοιραζόμαστε εκτιμήσεις για τις αμυντικές προσπάθειες Όμω όμως δεν έχει φτάσει ακόμη στο σημείο που θα θέλαμε να βρίσκεται η σχέση. Βεβαίως είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα πράγματα εδώ. Όμως, αν δούμε μόνο την ασφάλεια, θα δείτε ποιες είναι οι δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση κρίσεων και για την πολιτική παρέμβαση. Εκεί χρειάζεται βοήθεια οι Ηνωμένε Πολιτείε γιατί δεν έχουν τόσο αναπτυγμένες δυνατότητες. Αποτελεί προτεραιότητα αυτό για την κυβέρνηση Ομπάμα και έχουν έρθει οι ΙΠΑ στις Βρυξέλλες για να ρωτήσουν πώς μπορούμε να συνεργαστούμε επ' αυτό. Πάντως ε, σίγουρα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να αποφύγει και τις διάφορες θεολογικές συζητήσεις για τις σχέσεις ΕΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό γιατί το ΝΑΤΟ δεν ασχολείται τόσο με την ένωμη τάξη, με την καλή διακυβέρνηση, με την οικονομική ανικοδόμηση. Αυτά θα πρέπει να τα αναλάβουν η ΕΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι εταίροι. Αυτή τη στιγμή όμως δεν διαθέτουμε την κατάλληλη υποδομή, τις κατάλληλες δυνατότητες. Κοιτάξτε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανατολική σας πλευρά, στα ανατολικά σας σύνορα υπάρχουν πολλές αναταράξεις θεωρώ ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί κάποια εταιρική σχέση σε συνεργασία και με τις Ηνωμένε Πολιτείε για να προσπαθήσουμε να έχουμε σταθεροποίηση της κατάστασης εκεί όπως έχουμε κάνει και στα Βαλκάνια που παραμένει βασικό κομμάτι στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, για τις προτάσεις Μετβέντεφ, νομίζω ότι μας δίνουν μία δυνατότητα επί τη βάση των συμφωνιών του Ελσίνκη. Δηλαδή Ελσίνκη συν, όχι Ελσίνκη πλην. Πρέπει δηλαδή να ξεκινήσουμε με μία πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές του Ελσίνκη όπως το σεβασμό της ε, κυριαρχίας κάθε κράτους, της δυνατότητας κάθε κράτους να επιλέξει τους συμμάχους του και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι η ίδια με του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί έχουμε έναν κοινό στόχο, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, στην δεύτερη περίπτωση δεν μιλάμε για χώρες που έχουν κοινούς στόχους, αλλά μιλάμε για ένα κοινό πλαίσιο. Και αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να συνεχιστεί και να αξιοποιηθούν και προτάσεις όπως αυτού του κυρίου Μετβέντεφ. Για την ασφάλεια θεωρώ ότι αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ευρώπη προκλήσεις ευρείες που δεν νομίζω ότι τις έχουμε αντιμετωπίσει καλά που αφορούν την κοινωνία ασφάλειας. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την κυκλοφορία αγαθών, ανθρώπων, ενέργειας όλα αυτά στα οποία βασίζεται μια ελεύθερη κοινωνία, για όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι είτε από ανθρώπινες καταστροφές είτε όχι. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τις κατάλληλες δυνατότητες όλοι μαζί για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστροφικές προκλήσεις. Αυτό που είχε κάνει καλά ο ΑΣΕ μέχρι σήμερα ήταν να δώσει κάποιους κανόνες πορείας σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαφορές. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με αυτή την κοινωνία ασφαλείας και να βρούμε κάποιους βασικούς κανόνες για θέματα όπως την κυβερνοασφάλεια, την τρομοκρατία, την ενεργειακή ασφάλεια. Πρόκειται για θέματα που θα έπρεπε ο ΑΣΕ να λάβει σοβαρά υπόψη. Επίσης, όσον αφορά τις επιτόπου αποστολές του ΑΣΕ, είναι νομίζω το βασικό του δυνατό σημείο και πρέπει να εξακολουθήσουμε να τις τονίζουμε. Για παράδειγμα, Βοσνία. Γιατί πρέπει ο ΑΣΕ να αναλάβει το έργο της θεσμικής μεταρρύθμισης στη Βοσνία ρζεγοβίνη. Πρόκειται για θέμα θεμελιώδους σημασίας για αυτή την χώρα και νομίζω ότι η συμμετοχή του ΑΣΕ εκεί θα ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα. Επίσης, καθώς ε, εξακολουθούν να δημιουργούνται προκλήσεις στη Μεσόγειο, θα έπρεπε να αποκτήσει δυνατότητες ε, επίλυσης διαφορών και κρίσεων ο ΑΣΕ για να μπορεί να αποφύγει μελλοντικές κρίσεις. Τέλος, ας δούμε την συμφωνία για τα συμβατικά όπλα, η οποία μεταρρυθμίστηκε πρόσφατα αλλά δεν έχει επικυρωθεί από όλους και αποτελεί αυτή τη στιγμή εμπόδιο για την περαιτέρω πρόοδο. Η Ρωσία συμμορφώθηκε με κάποιες από τις προϋποθέσεις αλλά όχι όλες. Το ΝΑΤΟ δεν την έχει επικυρώσει, άρα βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο. Όμως αυτή η συνθήκη προσφέρει πολλά πλέον εκτήματα, με τον περιορισμό των όπλων και την δημιουργία κανόνων. Μας δίνει δηλαδή κάποια βασικά επίπεδα εμπιστοσύνης για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Νομίζω ότι το να μιλάμε για μελλοντικές συνθήκες είναι πρόημο. Πρέπει πρώτα να δούμε τι κάνουμε για να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις από τις Υπάρχουν συνθήκες. Άρα, συνοψίζοντας, επικροτώ τις προτάσεις Μετβέντεφ, αλλά η Ρωσία πρέπει να βρει πώς θα συμμορφωθεί πλήρως με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της στα πλαίσια της τελικής πράξης του Ελσίνκη. Και επίσης θεωρώ ότι η Δύση, ΝΑΤΟ αλλά και άλλοι οργανισμοί ήταν υπερβολικά παθητικοί για αυτή την πρόταση. Στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε ότι επικροτούν την πρόταση και θα υπάρξει διμερής διάλογος. Από τότε όμως σιωπή η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται γιατί από ό,τι φαίνεται είναι αμφίσιμη η σχέση της με τον ΟΑΣΕ. Κάποιες φορές αδιαφορεί, κάποιες φορές προσφέρει μόνο ρητορική βοήθεια, ορισμένες φορές προσπαθεί να ανταγωνιστεί τον ΟΑΣΕ. Για παράδειγμα Ευρωπαϊκή Αποστολή στην Γεωργία. Γιατί δεν ήταν αποστολή του ΟΑΣΕ αυτή, γιατί ήταν Ευρωπαϊκή Αποστολή, αφού αυτός ήταν ο λόγος δημιουργίας του ΟΑΣΕ. Οπότε σε ορισμένες περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΑΣΕ φαίνεται ότι συγκρούονται κατά κάποιο τρόπο, επικαλύπτονται. Πρέπει λοιπόν να δούμε Ποιε είναι οι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΑΣΕ και ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα παραμένει για πολλού ανθρώπου. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε και άλλους ομιλητές που θα πρέπει να παρέμβουν μετά τον πρώτο γύρο συζητήσεων. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσπαθήσετε να περιοριστείτε σε δύο λεπτά. Και θα ζητήσω από τους ομιλητές να απαντήσουν. Για να συνεχίσουμε με το δεύτερο γύρο. κύριος Βανόρντεν, παρακαλώ να παραμείνετε στα δύο λεπτά πολύ δύσκολο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές ε, Σιλβέστρη και Χάμιλτον για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Καταρχήν, σε σχέση με την ε, ιδέα της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ασφάλειας που ανέφερε ο πρόεδρος εξ αρχής, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχαμε στο παρελθόν ε, σοβιετικές βλέψεις και τώρα ρωσικές σε σχέση με μια ενδεχόμενη ενδεχόμενη, ε, ένα ενδεχόμενο σύμφωνο το οποίο θα απαγκίστρωνε την Ευρώπη από τις ΗΠΑ. Αυτό θα πρέπει να έχουμε πάντα. Είναι κάτι που θα πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου. ως προς την δημιουργία αυτής της ενδεχόμενης συνθήκης. Ως προς τα σχόλια του καθηγητού Σιλβέστρη το τελευταίο σημείο είναι και το πλέον σημαντικό. Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος έγκυται στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο σε θέματα άμυνας. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι παγκόσμιος φορέας με στρατιωτικές δυνάμεις για να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες της. Τη στιγμή που υπάρχει αυτό το πλαίσιο και τώρα έχει εγγραφεί και σε μία συνθήκη, εφόσον λοιπόν υφίσταται κάτι τέτοιο, υπάρχει μία ένταση στο ΝΑΤΟ, διότι τα περισσότερα μέλη είναι ευρωπαϊκές χώρες. Άρα δεν είναι ε, σίγουρες ε, το τι πρέπει να κάνουν. Δηλαδή δεσμεύονται ως προς το ΝΑΤΟ ή προσπαθούν να βρουν κάποιο ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεχωριστό ρόλο. Και οι επικρίσεις και οι αντιρρήσεις που ακούμε τώρα για την αναθεώρηση της στρατηγικής ε, έννοιας και συλλογιστικής έγκυται στο ότι δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αυτό επιθυμούν να δουν πολλοί. Μόνο όταν το ξεπεράσουμε αυτό θα λύσουμε το ζήτημα. Θα πρέπει να δούμε τις ε, φιλοδοξίες άμυνας για αυτό που είναι. Δηλαδή είναι πολιτικές βλέψεις, δεν είναι στρατιωτικές, ούτε έχουν σχέση με την στρατιωτική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν είμαστε πιο αποδυναμωμένοι διότι έχουμε κρατικές πολιτικές άμυνας. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θέλουν να ταχθούν υπέρ μιας ευρωπαϊκής, ευρωπαϊκής αρχής διότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν θέλουν μια ενιαία πολιτική άμυνας. Αυτό είναι και το πρωταρχικό μας μέλημα. Γιατί πολλοί μιλάνε για συζητήσεις δόγματος, για ζητήματα έμπρακτης εφαρμογής μέχρι ότου λυθεί αυτό το θέμα δόγματος όπου αναγνωρίζουμε ότι το ΝΑΤΟ είναι το στρατιωτικό σκέλος, μια στρατιωτική καθαρά οργάνωση η οποία αναπτύσσει τη στρατιωτική της ε, ικανότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να ασχοληθεί με τον πολιτικό τομέα, δηλαδή με το μη στρατιωτικό σκέλος. Πολλά μπορούν να λεχθούν επ' αυτού, αλλά αυτό είναι ένα θέμα ουσίας που ήθελα να θίξω. Η κυρία Γκόμες. Εγώ πιστεύω το αντίθετο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει αρκετά στον τομέα άμυνας και ασφάλειας και δεν είναι μόνο δικό μου ε, θέμα και άποψη. Το ζήτημα είναι ότι σε σχέση με την πολιτική Ομπάμα πώς μπορούμε εμείς να ανταποκριθούμε και να επιμερίσουμε αυτό το φόρτο διότι δεν μιλάμε για αντιμαχόμενες ε, δυνάμεις ή βλέψεις σε σχέση με τις ΗΠΑ, αλλά για ένα συμπληρωματικό χαρακτήρα. Πιστεύετε ότι η αναθεώρηση του στρατηγικού βασικού στόχου του ΝΑΤΟ αφορά σε μία αλλαγή ως προς το πυρηνικό δόγμα, δηλαδή σε στιγμές οικονομικής κρίσης μπορούν οι Ευρωπαίοι, δηλαδή ιδιαίτερα οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, να θέσουν κατά μέρος χρήματα στον τομέα των πυρηνικών Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει και πολιτική θέληση ως προς την τρομοκρατία που είναι μια άλλη απειλή όπου δεχόμαστε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή δόγματος. Δεν νομίζω ότι ήμασταν ε, αποτελεσματικοί ούτε από αυτή την πλευρά ούτε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δηλαδή, οι τρομοκράτες τι κάνουν, στρατολογούν μέλη Άρα υπάρχει θέμα πληροφόρησης, αντικατασκοπίας, κάτι στο οποίο εμείς οι Ευρωπαίοι δεν είμαστε πολύ καλοί. Υπάρχει το θέμα των κρατήσεων, όπου υπάρχουν αντικρουόμενες θέσεις και η κυβέρνηση Ομπάμα φοβούμε ότι εξακολουθεί να ε, αρκείται στις ίδιες θέσεις, δηλαδή ε, κάνει παράνομες κρατήσεις. Αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει κράτηση 48 προσώπων χωρίς να γίνεται δίκη. Άρα στην ουσία αυτά τα πρόσωπα μετατρέπονται σε μάρτυρες αντί για τορμοκράτες που είναι. Άρα δεν αντιμετωπίζουμε το θέμα των τρομοκρατών. Και δεν μιλώ μόνο για τη Μέση Ανατολή αλλά και για τη Σομαλία. για ότι στις ΙΠΑ οι τρομοκράτες οι περισσότεροι σχετίζονται με την Σομαλία. Έχουν κάποια διασύνδεση με τη Σομαλία και δεν κάνουμε ό,τι χρειάζεται σε αυτό το τομέα. Κύριε Κοπά. Πρόεδρε, ε, διαβάζοντας το κείμενο της ομάδας των σοφών θα μπορούσα να συγκρατήσω τέσσερα σημεία. Πρώτα απ' όλα την ανάγκη να απαντηθεί το υπαρξιακό ερώτημα για τους λόγους ύπαρξης του νατο μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και τη μετά της 11 η σεπτεμβρίου εποχή. Δύο, τη δέσμευση για μια αναθεώρηση του άρθρου 5 αλλά και τη διεύρυνση των προϋποθέσεων ε, ε, εφαρμογής τους την διερεύνηση μάλλον των νέων προϋποθέσεων για την εφαρμογή τους ε, τρία την προσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα σε αποτελεσματική αποτροπή και μείωση στο ελάχιστο των πυρηνικών όπλων στη συμμαχία και τέταρτον την επιδίωξη στενότερης συνεργασίας με τη ρωσία. Ε, η νέα, το νέο στρατηγικό δόγμα του νάτο θα κριθεί εκτός των άλλων αλλά κατά πολύ βασικό τρόπο στην περίπτωση του αφγανιστάν. το νάτο συνεχίζει μαζικά την παρουσία του εκεί και δύο θα είναι τα κρίσιμα ερωτήματα. Πρώτον, αν ε, μπορεί στη βάση μιας ενδεχόμενης επιτυχίας, που είναι πολύ αβέβαιη αυτή τη στιγμή, να αναλάβει άλλες επιχειρήσεις σε ε, εξωτερικές περιοχές, σε άλλες περιοχές στο μέλλον και δεύτερον, αν μπορεί να λειτουργήσει η ε, επωνομαζόμενη ενιαία πολιτικοστρατιωτική προσέγγιση, το comprehensive approach, με συνδυασμό στρατιωτικών και πολιτικών μέσων. Ε, πολύ ενδιαφέρον στο κείμενο είναι η αναγνώριση στο σημαντικό ρόλο της Ρωσίας για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος ασφαλείας στην ευρύτερη ευρασιατική περιοχή. Όμως το κείμενο δεν προχωράει σε ουσιαστικές προτάσεις για την ενδυνάμωση της εταιρική σχέσης. Αναφέρει ότι η πόρτα είναι ανοιχτή σε όλα τα επίπεδα, χωρίς όμως να εξειδικεύει, περιοριζόμενο στην παρούσα δομή συνεργασίας του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι ε, πώς μπορούμε να φανταστούμε νέους αποτελεσματικότερους μηχανισμούς συνεργασία με τη Ρωσία. Και μια και ε, θα συζητήσουμε και το θέμα του ΟΑΣΕ, ίσως θα μπορούσε να αναφερθεί αυτός ο οργανισμός στο κείμενο, κείμενο σαν ένα διάβλο ε, συνεργασίας μεταξύ Ανατολής και Δύση και ειδικά ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και στη Ρωσία. Ε, Πάντως υποθέτω και σε αυτό θα ήθελα τη γνώμη σας ότι αυτό το κείμενο φυσικά δεν είναι δεσμευτικό, υπάρχουν δυνατότητες για αλλαγές και προς ποια κατεύθυνση θα βλέπατε εσείς αυτές τις ενδεχόμενες αλλαγές μέχρι τον Νοέμβρη. Ευχαριστώ. Thank you very much. Mrs. Lösing, please. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κυρία Λέζινγκ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σιλβέστρη, Είπατε ότι αναμένεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εμβαθύνει την αμυντική της στρατηγική. Τι εννοείται εμβαθύνει. Η εντύπωση μου είναι ότι έχει δύο πτυχές. Αφενός να επεκταθεί η έννοια της ασφάλειας και αφετέρου να αυξηθούν οι δαπάνες εξοπλισμών. Αυτά πάνω στον καμβά της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, όπου λαμβάνονται παντού μέτρα εξοικονομήσεων, όπου οι άνθρωποι βλέπουν να καταραίουν τα κοινωνικά συστήματα ασφάλισης. Και μέσα σε αυτή την περίοδο κρίσης ζητάτε αυξήσεις των στρατιωτικών εξοπλισμών. Στην έκθεση ΝΑΤΟ 2020 που συντάσσει η Επιτροπή που έχει ορίσει ο Γενικό Γραμματέας του ΝΑΤΟ ζητιέται ξεκάθαρα από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να προβούν σε υψηλότερε αμυντικές δαπάνες για να προωθήσουν την συνεργασία με τις ΗΠΑ. Συμφωνείτε με την εκτίμηση αυτή. Στην ομιλία σας και στην έκθεσή σας για την ISS European Defense είπατε να, να μπουν κάποιες ημερομηνίες και κάποια ε, μέχρι τις οποίες να γίνουν οι αυξήσει αυτές, αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία. Έχετε συγκεκριμένα, έχετε συγκεκριμένα τέτοια δεδομένα και ποια είναι αυτά. Το θέμα του ΟΑΣΕ και της συμπερίληψης της Ρωσίας θα ήθελα να το θέσω στον επόμενο γύρο ερωτήσεων. Όταν όμως στις δημοσκοπήσεις ρωτούν τους πολίτες μας στους δρόμους τι φοβούνται, ο φόβος που εκφράζουν είναι μη χάσουν τις δουλειές τους. Δεν φοβούνται εξωτερικές απειλές. Η φτώχεια είναι αποδεδειγμένο ότι είναι η νούμερο ένα παγκόσμια αιτία που οδηγεί σε συγκρούσεις. Και τέλος για το πρόβλημα της τρομοκρατίας. Ναι, πολλοί άνθρωποι φοβούνται την τρομοκρατία, αλλά και εδώ εγώ επιθυμώ να ξεκαθαρίσω ότι η συμμετοχή των χωρών σε πολεμικές επιχειρήσεις ε, στο εξωτερικό οδηγεί πάλι σε αντίδραση των τρομοκρατών και εγώ θεωρώ ότι πάλι διασυνδέεται εκεί η φτώχεια με την τρομοκρατία. Ο κύριος Αγκουράκης παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δύο παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα μου έκανε μεγάλη εντύπωση στην ε, τοποθέτηση του καθηγητού Χάμιλτον εγώ τουλάχιστον για πρώτη φορά τα ακούω, στους λόγους ύπαρξης του ΝΑΤΟ, ο αξιότιμος καθηγητής αναφέρθηκε και στην ασφάλεια που νιώθουν οι ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ τους. Αν κατάλαβα καλά και αν ήταν σωστή η ελληνική μετάφραση, ότι το ΝΑΤΟ τους παίρνει τον φόβο του ενός από τον άλλο. δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά. Αν κατάλαβα καλά, αυτό με οδηγεί στο να σκεφτώ ότι και ο κύριος καθηγητής σκέφτομαι όπως και εγώ περίπου ότι δυστυχώς λόγω της ανάπτυξης της κρίσης και λόγω των υπεριαλιστικών χαρακτηριστικών των σύγχρονων καπιταλιστικών χωρών οδηγούμαστε σε μια περίοδο που εμένα μου θυμίζει λίγο την παραμονή του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Και το λέω αυτό κύριε καθηγητά μου διότι κατά τη γνώμη μου το μόνο καινούριο πραγματικά στοιχείο που υπάρχει να σας κάνει, να κάνει την κυβέρνησή σας και τις κυβερνήσεις των χωρών μελών του ΝΑΤΟ να συζητάνε μια νέα στρατηγική του ΝΑΤΟ μετά από την προηγούμενη αναθεώρηση είναι πρώτον ο μεγάλος ανταγωνισμός για τα ενεργειακά και κακά τα ψέματα εδώ δεν έγινε καμία συζήτηση αλλά ξέρουμε πόσο μεγάλος είναι αυτός ο ανταγωνισμός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ηνωμένε Πολιτείε με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της ενέργειας και δεύτερον είναι η μεγάλη αποτυχία της επιχείρησης στο Αφγανιστάν γι' αυτό κιόλας και η κυρία Όλμπραϊτ και οι πολιτικοί ε, ηγέτες του ΝΑΤΟ μιλάνε ότι το Αφγανιστάν είναι το κλειδί για το μέλλον του ΝΑΤΟ. Και η ερώτηση μου είναι η κύριε καθηγητά Το είπε και η κυρία Κοπά πριν ένας από τους λόγους της νέας στρατηγικής είναι το άρθρο 5 της Συμμαχίας. Το άρθρο 5 της Συμμαχίας, αγαπητέ μου κύριε καθηγητά, προβλέπει η εφαρμογή του μόνο σε, μόνο σε περίπτωση επίθεσης στο έδαφος των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Αυτός είναι και ο λόγος εξάλλου που μετά τις 11 Σεπτεμβρίου ο κύριος Ράμσφελτ δεν μπόρεσε να επικαλεστεί το άρθρο 5 και μίλησε για μια συμμαχία των προδήμων στο Αφγανιστάν. Εσείς θέλετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω εγώ ποιο, ή η ομάδα των ε, ε, σοφών, το άρθρο 5 να ισχύει ακόμα και σε περιπτώσεις για επιχειρήσεις σε οποιαδήποτε σημείο του κόσμου. Γι' αυτό το λόγο... Τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω την άποψή για το ζήτημα αυτό. Έχουμε στον κατάλογο τον κύριο Μπουτικόφερ και τον κύριο Λαντσπέργης. Αλλά επειδή θα θέλαμε να συνοψίσουμε αυτή τη συζήτηση εγκαίρως, πριν από την επόμενη συζήτηση, θα ήθελα να ζητήσω από τις δύο άλλες ομιλήτριες να λάβουν το λόγο και μετά θα ε, συνεχίσουμε. Θα έχουμε δηλαδή μία σύντομη απάντηση από τους κυρίους, θα μιλήσουν οι κυρίες και μετά θα ανοίξει η συζήτηση. Οι κύριοι θα παραμείνουν και θα είναι σε θέση να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας. Γίνεται μία μικρή ανατροπή, αλλά θα ήθελα να μιλήσουν και οι κυρίες, να έχουν το χρόνο. Λοιπόν, θα ήθελα ο, η Στέφανο και Ντάνιλ να απαντήσουν εν συντομία και μετά θα λάβουν το λόγο οι κυρίες. Προς τον κύριο Βανόρτεν, θα ήθελα να πω ότι κατά την άποψή μου το ΝΑΤΟ θα πρέπει να επιλύσει το θέμα της συλλογική ασφάλειας. Δυστυχώς, αν λάβουμε υπόψη την παρούσα κατάσταση της απειλής και επειδή δεν μπορεί να αναγνωριστεί πλήρως και μεταλλάσσεται, πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη συλλογική ασφάλεια. Διότι υπάρχει μια εξελικτική πορεία για την Συμμαχία των Προθήμων, για τις δράσεις της Συμμαχίας των Προθήμων. Και αυτό αποδυναμώνει την αλληλεγγύη μεταξύ των συμμάχων. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, αλλά βλέπετε ότι ως προς την απειλή υπάρχουν δύο ή τρεις ομάδες συμμάχων, δηλαδή μια διαφορετική οπτική γωνία της απειλής. Συμφωνώ με τον συνάδελφο ε, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η συμμαχία είναι άχρηστη, αλλά δεν είναι η ίδια με αυτή που υπήρχε κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και δεν διαδραματίζει τον ίδιο ρόλο. Όταν μιλάμε για στρατιωτική δράση ή πολιτική δράση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουμε έναν διαχωρισμό που έρχεται σε αντίθεση με τη συνεκτική αυτή προσέγγιση. Προς την κυρία Γκόμες θα ήθελα να πω ότι κατά την άποψή μου οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να δαπανούν ε, λίγο περισσότερο σε θέματα άμυνας, όχι πολλά, όχι πολύ περισσότερο, διότι θεωρήσαμε ότι οι Ευρωπαίοι θα δαπανούν ένα 2% μέσο όρο του ΑΕΠ. Τώρα βρισκόμαστε στο 1% μέσο όρο και ίσως και λιγότερο. Αν θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούμε στη νέα αυτή κατάσταση, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια αναθεώρηση ως προς τη χρήση των πυρηνικών από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, η οποία θα αντιστάθμιζε την κατάσταση. Θα πρέπει να γίνει καλύτερος τρόπος δαπάνησης και θα πρέπει να μειωθεί ο κατακαιρματισμός της δαπάνης που έχει καθαρά εθνικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι οι δαπάνες θα πρέπει να οργανωθούν ως εξής. Ως προς τους στρατιωτικούς σκοπούς θα πρέπει να αποφασίζονται από μερικές χώρες αποκλειστικά και είναι γεγονός ότι τέσσερις ή πέντε χώρες, μάλλον επτά χώρες αποτελούν σχεδόν το σύνολο των αμυντικών δαπανών. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά τον προγραμματισμό. Δεν είναι αναγκαία κάτι το καλό. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει κοινός προϋπολογισμός. Είναι κάτι που θα πρέπει να εξελιχθεί, αλλά δεν υπάρχει ακόμα. ως προς την ε, συμμετοχή στις πληροφορίες, στην αντικατασκοπία, δεν ξέρω ε, ότι έχει αναπτυχθεί επαρκώς αυτό το σκέλος. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ζήτηματα κρίσης, όπως η νέα κρίση που αντιμετωπίζουμε. Προς την κυρία Κοπά, θα ήθελα να πω ότι όλοι όσοι πιστεύουν ότι το άρθρο 5 μπορεί να διευρυνθεί ή να επανερμηνευθεί, ε, νομίζω ότι αυταπατώνται. Διότι το άρθρο 5 ήταν ένας πολύ δύσκολος συμβιβασμός. Μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά, μπορεί να το πει κανείς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι νομικά μπορείτε να το αλλάξετε. Είναι γεγονός ότι αν αρχίσουμε να επανασυζητούμε το άρθρο 5 θα τελειώσουμε με το ΝΑΤΟ και θα έχουμε μια πολύ δύσκολη θέση με τις ΙΠΑ. Θα ήταν πολύ καλύτερα να αρχίσουμε με μια διαδικασία διαβουλεύσεων σε θέματα άμυνας μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ για να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές προτεραιότητες σε, στις περιφέρειες μεγαλύτερου ενδιαφέροντος, μίζωνος ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αυτό δεν το έχει αποσαφηνίσει κανείς. Και εδώ έχουμε δύο φορείς, δύο χώρες που είναι πολύ σημαντικές, που έχουν διαφορετικές θεωρήσεις του ρόλου των ΙΠΑ. Είναι η Ρωσία και η Τουρκία. Ως προς άλλες παρατηρήσεις δεν έχω και πολλά να πω. Συμφωνώ ότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες περί άμυνας, γιατί εγώ για άμυνα μίλησα αποκλειστικά. Και βεβαίως είναι ένα θέμα πολιτικών αποφάσεων και προτεραιοτήτων. Κατά την άποψή μου, είναι δυνατόν να έχουμε μία αποτελεσματική άμυνα χωρίς να παρεμποδίσουμε την οικονομική ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Και εγώ πιστεύω ότι το άρθρο 5 θα πρέπει να παραμείνει ως έχει, γιατί είναι θέμα ε, καθαρά ε, Μετά την, ε, ε, την τρομοκρατική δράση της 11 η Σεπτεμβρίου, ερμηνεύσαμε αυτό το άρθρο. Άρα γιατί να μην ε, συνεχίσουμε σε αυτή την οδό, κύριος Βανόρτε. Ένα θέμα διασάφησης, κύριε Πρόεδρε, διότι ο καθηγητής Σιλβέστρη αναφέρθηκε σε μια συνολική προσέγγιση, σαν να τάσετε κατά της εξειδίκευσης ρόλων. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι δεν ισχύει δεν υπάρχει τίποτα το καινούριο ως προς την συνολική προσέγγιση. Δηλαδή μιλάμε με την καρδιά και με το νου. Κανένας στρατιώτης δεν θεωρεί ότι μπορεί να κερδίσει μόνο με στρατιωτικά μέσα. Ε, όλοι πιστεύουν στο δόγμα του Φον Κλάουζοβιτς. Δηλαδή χρησιμοποιούν τον χώρο έτσι ώστε να μπορέσουν να δράσουν Άλλη, Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θέλει να κάνει και τα δύο. Θέλει να δράσει και στο στρατιωτικό και στο πολιτικό σκέλος. Και αυτό υποβαθμίζει την θέληση των συμμάχων να επιτύχουν στο Αφγανιστάν. Διότι δεν υποστηρίζουν αυτή τη δράση όπως θα έπρεπε. Ας μην θεωρήσουμε λοιπόν ότι η συνολική προσέγγιση σημαίνει ότι όλα τα βάζουμε σε ένα κουτί. Χρειάζεται συντονισμός μεταξύ στρατιωτικής και μη στρατιωτικής δραστηριότητας, αλλά αυτό δεν τάσεται κατά της εξειδίκευσης ρόλων και δραστηριοτήτων. Συμφωνώ με αυτό και έτσι υποθέτω ότι απαντώ στο πρώτο ερώτημα. Ένα δεύτερο ερώτημα όσον αφορά την αλλαγή του ποινικού δόγματος. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιου είδου προσπάθειες αυτή τη στιγμή. Συνήθως μιλάμε για την σημασία της, ε, της αποφυγής, ε, της ε, απόπισης Νομίζω ότι αυτό το θέμα ίσως ε, διαφορετικά ε, έχει διαφορετική σημασία για τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δείτε τις τελευταίες πυρηνικές προσπάθειες, θα δείτε ότι δεν προσπαθήσαμε να πιέσουμε τους Ευρωπαίους. Αν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή άποψη ότι δεν είναι απαραίτητα αυτά τα πυρηνικά όπλα, θα τα ή, θα τα είχαν αποσύρει οι Ηνωμένε Πολιτείε. Όμως δεν νομίζω ότι υπάρχει ευρωπαϊκή άποψη, δεν υπάρχει συνένεση για αυτό το θέμα στην Ευρώπη και γι' αυτό παραμένουν. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της Συνόδου. Τώρα όσον αφορά το άρθρο 5 και την διασφάλιση των Ευρωπαίων. Κοιτάξτε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και για το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, οι ευρωπαϊκοί στρατοί κατευθύνονταν ο ένας εναντίον του άλλου και μετά την μεγάλη τραγωδία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου ξεκίνησαν να συνεργάζονται. Αυτή τη στιγμή Γάλλοι και Γερμανοί δεν ε, δημιουργούν αμυντικές ε, δυνατότητες για να καταπολεμήσουν ο ένας τον άλλον. Αυτή τη στιγμή Ελλάδα και Τουρκία δεν έχουν πολύ καλές σχέσεις, αλλά εντός του ΝΑΤΟ έχουν καταφέρει να μην οδηγηθούν σε σύραξη. Άρα Υπάρχει αυτή η διασφάλιση από την συμμαχία του ΝΑΤΟ που ορισμένες φορές ε, την ε, παραβλέπουμε. Θα σας ρωτούσα πραγματικά, θεωρείτε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι αρκετή, θεωρείτε ότι αν δεν υπήρχε το ΝΑΤΟ θα αισθάνοσταν άνετα για την ασφάλειά σας. Είναι ένα βασικό ερώτημα αυτό και πιστεύω ότι παραμένει αυτός ο ρόλος του ΝΑΤΟ ακόμη και καθώς αναπτύσσεται όλο και περισσότερο η Ευρώπη. Τώρα, το ερώτημα για τη διεύρυνση του άρθρου 5 και για την 11η Σεπτεμβρίου δεν νομίζω ότι το κατάλαβα καλά. Η Νέα Υόρκη και η Ουάσιγκτον είναι κομμάτι της περιοχής του χώρου δράσεως στο ΝΑΤΟ. Δεν υπήρξε προσπάθεια επέκτασης του γεωγραφικού χώρου. Είναι κομμάτι ιστορικό. Άρα αν μιλάμε τώρα για επέκταση του άρθρου 5, εγώ όντως θα έλεγα ότι αυτό είναι υπερβολικός στόχος. Όμως αυτό που βλέπω σήμερα είναι μεγαλύτερη σημασία για το άρθρο 4. Αυτό το βλέπετε και στην έκθεση των σοφών, οι οποίοι τονίζουν τη σημασία να έχει καλύτερες εταιρικές σχέσεις στο ΝΑΤΟ να έχει καλύτερες συνεργασίες γιατί αυτή τη στιγμή δεν τα πάει τόσο καλά σε αυτό το τομέα αλλά θα πρέπει να το επιτύχει αυτό για το μέλλον. Πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τις εταιρικές σχέσεις να κάνει συμμαχίες. Και όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 4. Και εκεί συμπεριλαμβάνονται και οι εταιρικές σχέσεις για την ειρήνη, τα Partnership for Peace Και νομίζω ότι μετά τη Σύνοδο της Λισαβόνας το άρθρο 4 θα είναι ακόμη πιο σημαντικό. Επίσης, συμφωνώ με αυτό που αναφέρθηκε ότι το ΝΑΤΟ σήμερα δεν επαρκεί για τις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε. Είναι σημαντικό, αλλά είναι και ανεπαρκές, γιατί δεν έχει όλα τα εργαλεία που χρειαζόμαστε. Όμως θα πρότεινα κάτι διαφορετικό. Αντί να επεκτείνουμε το άρθρο 5, που δεν θα σήμαινε και τίποτα, να κάνουμε λίγο πίσω και να σκεφτούμε όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα και ενδεχομένως να καταλήξουμε σε ένα διαφορετικό συμπέρασμα. Η μοναδική υποχρέωσή μας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού είναι το άρθρο 5. Απάντηση σε ένοπλη επίθεση. Όμως, οι απειλές για τις οποίες μιλάω τώρα ενδεχομένως δεν είναι ένοπλες επιθέσεις. Μπορεί όμως να είναι πολύ πιο πραγματικές απειλές για την ασφάλεια ενός κράτους. Οπότε, ίσως θα έπρεπε να επεκτείνουμε αυτό που σήμερα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση καταστροφής θα βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Γιατί να μην το πούμε αυτό. Για να μην υπάρξει μια δέσμευση αλληλεγγύης βορειοατλαντική που θα συμπληρώνει το πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Κάτι διαφορετικό δηλαδή, κάποια πολιτική αλληλεγγύη. Το ίδιο που κάνουμε και τώρα με τον κόλπο του Μεξικό, που χρειαζόμαστε ενδεχομένως το ίδιο πρόβλημα που είχαμε και με τον τυφώνα Κατρίνα όπου μας βοήθησε ο υπόλοιπος κόσμος παρόλο που θεωρούσαμε ότι δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Αυτά είναι παραδείγματα αλληλεγγύης και ενδεχομένως, αν και το απέφχομαι, να χρειαστεί και εμείς να βοηθήσουμε την Ευρώπη σε μια φυσική άλλη καταστροφή. Άρα, θα έπρεπε να δούμε και με αυτές τις διαστάσεις της ασφάλειας την σχέση είπα και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τρύπα, ένα κενό στην αρχιτεκτονική ασφαλείας που δεν έχει αναπτυχθεί όσο θα έπρεπε. Uh, Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην πρέσβυρα κυρία Μαρινάκη και στη δόκτωρα Αρπάτοβα για να μιλήσουν για την μεταρρύθμιση ΟΑΣΕ και για την πρόταση Μετβέντεφ για μια ευρωπαϊκή συμφωνία ασφάλειας και μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τους κύριους Μπούτικοφ και Λαντσβέργης καταρχάς. Είναι μεγάλη τιμή για μένα κύριε Πρόεδρε να βρίσκομαι εδώ σήμερα μπροστά σας για να συζητήσω για ένα θέμα το οποίο απασχολεί τα τελευταία χρόνια την ευρωατλαντική εταιρική σχέση. Με λίγα λόγια, θα σας εξηγήσω ποιες είναι οι βάσεις της εμπειρίας μας για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας της Κέρκυρας που έρχεται και μετά από την Προεδρία του ΟΑΣΕ στην, ε, το 2009 μετά από τεράστιες προκλήσεις για την ευρωθρατική ε, ασφάλεια. Η κρίση έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν το εφαλτήριο για βελτιώσεις και πράγματι η κρίση του 2008 και η σύγκρουση στην Γεωργία άλλαξαν τις ιδέες μας περί της ασφάλειας στην περιοχή εκείνη. Το 2009 ήταν βέβαια και η 20 ετία από την πτώση του τείχους του Βερολίνου και από το τέλος του ψυχρού πολέμου. Επέτειος και εορτής και αναλογισμού του, της πρόοδου που κάναμε τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά και στοχασμού για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Η κρίση του 2008 κατέστησε σαφές ότι το όραμα μιας ενωμένης Ευρώπης βασισμένης σε κοινέ αρχές και σε μια διαίρετη ασφάλεια που τόσο εύγλωτα είχε ε, διατυπωθεί στην τελική πράξη του Ελσίνκη του 1975 και στην πράξη των Παρισιών ακόμα δεν είχε υλοποιηθεί για όλους τους λόγους της Ευρώπης. Το όραμα παραμένει ένα στόχος ακόμα για ορισμένους. Η βασική διαφορά μεταξύ του Δεκεμβρίου 2008 και Δεκεμβρίου 2009 είναι ότι εν τω μεταξύ και οι 56 χώρες που συμμετέχουν στον ΟΑΣΕ επανεπιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους συνεργασίας για να επιτύχουν το όραμα αυτό στην βάση του κεκτημένου του ΟΑΣΕ και για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε, συμμετέχουμε όλοι στην ε, σκέψη αυτή να έρθω σε ορισμένα από τα στοιχεία του εγγράφου του ΟΑΣΕ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Πρώτο, ο δεκάλογος του Ελσίνκη με τις βασικές του αρχές διασύνδεσης της διακρατικής ασφάλειας με την ενδοκρατική σταθερότητα. Συνολική προσέγγιση προς την ασφάλεια βασισμένη στην βασική αρχή ότι η ασφάλεια είναι αδιέρετη, όπως λέει και η Χάρτα των Παρισιών του 1990. Η ασφάλεια είναι αδιέρετη και η ασφάλεια κάθε συμμετέχουσας χώρας διασυνδέεται με την ε, ασφάλεια όλων των υπολείπων. Το 1999, στο χάρτη της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας, ο ΑΣΕ Κωνσταντινούπολη, ε, όπου οι συμμετέχουσες χώρες επανέλαβαν τη δεσμευσή τους ότι θα δημιουργήσουν σχέσεις βασισμένες σε κοινή αρχή αδιέρετης ασφάλειας βασισμένη σε εταιρική σχέση, αλληλεγγύη και διαφάνεια. Η ασφάλεια της κάθε συμμετέχουσας χώρας ε, συνδέεται άρρηκτα. Παρακαλώ λίγο πιο σιγά. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο που επεσήμανε στην ομιλία του να μιλάει λίγο πιο αργά. Η στρατιωτική ή πολιτική διάσταση λοιπόν της ασφάλειας. Μετά το 1994 ο κώδικας διοντολογίας για τα πολιτικοστρατιωτικά που λέει επίσης ότι οι χώρες μέλη δεν θα ενισχύσουν την ασφάλειά τους σε βάρος της ασφάλειας άλλων χωρών. Και οι 56 λοιπόν χώρες που συμμετέχουν στον ΑΣΕ επετέλεσαν τα καθήκοντα αυτά. Νομίζω όχι. Οι περισσότερε από τις αρχές αυτές είτε παραβιάστηκαν, είτε ερμηνεύτηκαν εσφαλμένα, είτε εφαρμόστηκαν ε, επιλεκτικά. Το Ιανουάριο του 1900 του 2009 μάλλον, όταν ανέλαβε την Προεδρία η Ελλάδα, αμφισβητούνταν σχεδόν όλα τα ε, στοιχεία του χάρτη. Ανεπίλητες μεθοριακές ε, διαφορές, συγκρούσεις στον Κάφκασο και στην Ανατολική Ευρώπη, διακοπή δημοκρατικών διαδικασιών σε τμήματα της περιοχής του ΑΣΕ, και εκκρεμής ο μηχανισμός δημιουργίας ε, CFE δηλαδή για έναν αριθμό ετών που υποτίθεται ότι είναι και θεμελιώδες στοιχείο η e e. Αυτή η προσπάθεια αφοπλισμού έχει οδηγήσει στην κατάργηση 60.000 ε, τμήματων ε, βαρέων όπλων. Το πιο σοβαρό, οι εντάσεις και η δυσπιστία μεταξύ χωρών στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιφέρεια έχουν υποσκάψει την ε, ε, κοινή αντιμετώπιση και στο Αφγανιστάν και αλλού. Πολλοί λοιπόν θεώρησαν ότι η προσπάθεια αυτή είχε φτάσει σε ένα τέλος και το είχαν θεωρήσει αυτό και στην Ανατολική και στην Δυτική Ευρώπη. Η ο πρώτος κόδων κινδύνου ήταν το 2008 όταν ο πρόεδρος Μεντιέντεφ της Ρωσίας ζήτησε να υπάρξει διάλογος για την ε, βελτίωση των μηχανισμών ασφάλειας της Ευρώπης. Εάν τώρα η Ρωσία θεωρεί δίκαια ή άδικα ότι δεν αντιμετωπίζεται ως ισότιμος εταίρος στο σύστημα ασφάλειας της Ευρώπης, αυτό οφείλει να θεωρηθεί ως σοβαρό πρόβλημα, όχι μόνο για τη Ρωσία, αλλά για όλα τα μέλη της κοινότητας του ΟΑΣΕ. Το νόημα της ε, ε, έκκλησης αυτής της Ρωσίας αναγνωρίστηκε από τον πρόεδρο Σαρκοζή, ο οποίος ζήτησε να υπάρξει μια κοινή προσέγγιση και αυτό να αποτελέσει πηγή έμπνευση για όλες τις χώρες του ΟΑΣΕ να αφιερώσουν χρόνο και προσπάθεια ώστε να υπάρξει σιγά σιγά μια σταδιακή βελτίωση της ε, ασφάλειας. Από την αρχή η ελληνική προεδρία θεώρησε ότι οι προκλήσεις αυτές πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως εφαλτήριο για να ε, υπάρξει μια προσπάθεια διόρθωσης της κατάστασης. Επίσης θεωρούσαμε εμείς ότι ένας καλόπιστος και ανοιχτός διάλογος έπρεπε οπωσδήποτε να διεξαχθεί για τις μελλοντικέ προκλήσεις στην περιοχή του ΟΑΣΕ. Τώρα οι φάσεις της διαδικασίας της Κέρκυρας από Τελσίνκη μέχρι την Κέρκυρα αρχίσαν οι πρώτες ανταλλαγές απόψεων το 2008 από το στάδιο εκείνο, στο στάδιο εκείνο υπήρχαν περισσότερε ερωτήσει από απαντήσει. Μετά από ένα εξάμεινο και μετά από διαβουλεύσει στην Βιέννη, οι 56 υπουργοί συναντήθηκαν ξανά τον Ιούνιο του 2009, πάλι στην Κέρκυρα, όπου συμφώνησαν επί τη ανάγκη να εξετάσουν όλοι μαζί τι προκλήσει τη ασφάλεια στην Ευρώπη και τη ασφάλεια τη Ευρώπη, ένα πνεύμα συνεργασία και μέσα στα πλαίσια του κεκτημένου του ΟΑΣΕ αποφάσισαν δύο πράγματα βασισμένοι στις κατευθείαν γραμμέ που κρίθηκαν στην ΟΑΣΕ οι 56 αποφάσισαν να κάνουν ε, συζητήσεις για να αναπτύξουν μια κοινή ερμηνεία του ποιε είναι κατά προτεραιότητα οι προκλήσει στην ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια. Στη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, η διαδικασία τη Κέρκυρα άρχισε να αποδίδει του πρώτου καρπού τη μέσα σε πλαίσια αμοιβαίου σεβασμού, γενικής προθυμίας να ακούσουν οι μεν τους δε, καλύτερη κατανόησης και βελτίωσης σταδιακά του πνεύματος συνεργασίας. Αλλά πιο σημαντικό, άνοιξε τον δρόμο για την έγκριση της πολιτικής διακήρυξης της Κέρκυρας που έγινε στην Αθήνα. Έτσι η διαδικασία της Κέρκυρας που ξεκίνησε ως πρωτοβουλία της Προεδρίας έγινε τελικά το κοινό προϊόν της προσπάθειας των 56 χωρών. Δεν θα ήταν όμως πλήρης η προσπάθεια εάν δεν είχε περιλάβει και την κοινοβουλευτική συνέλευση. Έτσι λοιπόν στην Υπουργική Διέσκεψη της Αθήνας τον Δεκέμβριο οι Υπουργοί αποφάσισαν να προσκαλέσουν την κοινοβουλευτική συνέλευση καθώς και τους εταίρους της Μεσογείου και της Ασίας για να συμμετάσχουν στις προσπάθειες αυτές. Από την Αθήνα τώρα στο, στην Αλμαμάτα του Καζακστάν ακολούθησε η ε, Προεδρία του Καζακστάν με συγκεκριμένες προτάσεις για την βελτίωση σε όλους τους τομείς των ικανοτήτων του ΑΣΕ, όπου δηλαδή είχαν διαπιστωθεί ε, ελλείψεις. Αυτές τώρα συζητούνται και το πιο σημαντικό ακόμη είναι ότι μέσω διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών βαθαίνει η αμοιβαία κατανόηση και αναλαμβάνονται βαθύτερα οι δεσμεύσει. Η αξία τη διαδικασία εγγύεται στην ίδια τη διαδικασία. Α μην λησμονούμε ότι στα πλαίσια τη διαδικασία του Ελσίνκη πριν από 35 χρόνια παραπάνω από 4.600 προτάσει, έχουν κατατεθεί και συζητηθεί πριν από την έγκριση τη τελική πράξη του Ελσίνκη. Και μέσω των ανταλλαγών αυτών αναπτύχθηκε το πνεύμα του Ελσίνκη και οδήγησε εν τέλει στην επανένωση της Υπήρου Τώρα, προς τα πού θα κινηθούμε από εδώ. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η εξομάλυνση των διαφορών, η επανάκτηση της ε, κοινότητας των στόχων χρειάζεται χρόνο. Η επίλυση των ε, προβλημάτων της ε, Ευρώπης χρειάζεται κάτι παραπάνω από μια καλή ατμόσφαιρα. Χρειάζεται λοιπόν ένα μείγμα ρεαλισμού και φιλοδοξίας με αναζήτηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων παρόλο που μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από ό,τι υπολογίζεται ήταν στην αρχή. Έτσι λοιπόν στην Άλμα Μάτα στις 16 και 17 Ιουλίου η συνδιάσκεψη των Υπουργών εκεί θα δώσει περαιτέρω κατευθύνσεις για την ενίσχυση της διαδικασίας με υψηλότερους, φιλοδοξότερους στόχους μεταξύ του, της Μάτα και την Αστανά που θα γίνει στα τέλη του χρόνου. Ταυτόχρονα είμαστε πεπισμένοι ότι η διάσκεψη κορυφής της Αστανά δεν θα σημάνει το τέλος του δρόμου. Βρισκόμαστε μόνο στην αρχή του τέλους της διαδικασίας της Κέρκυρας. Παραπέρα, όπως προτείνει η Προεδρία του Καζακστάν, θεωρούμε ότι χρειάζεται να διατηρήσουμε αυτή την ορμή που έδωσε η επικοδομητική ορμή που έδωσε η ε, διαδικασία της Κέρκυρας για στρατηγικούς στόχους για μια συνολικότερη αντιμετώπιση της ασφάλειας σε ένα πιο δομημένο πλαίσιο. Μια ένα στρατηγικό όραμα λοιπόν αρχίζει και βρίσκει μεγαλύτερη υποστήριξη μια σύγχρονη συνεργασία από το Βανκούβερ μέχρι το Βλαδιβοστόκ, όπου κανένα δεν θα θεωρεί ότι μένει απ' έξω ή ότι παραγωνίζεται, όπου η χρήση βία δεν θα αποτελεί πλέον επιλογή. Κυρίε και κύριοι, μια ερώτηση που ακούγεται συχνά είναι γιατί ο διάλογο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια να γίνεται στο ΟΑΣΕ και όχι σε κάποιο άλλο βήμα. Δύο βασικοί λόγοι Πρώτον, η συμμετοχή στον ΟΑΣΕ ολόκληρου του Βόρειου Ημισφαιρίου σε ισότιμη βάση όλων των ενδιαφερομένων ορών για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και δεύτερον η βασική αρχή της ΟΑΣΕ μιας αδιέρετης και ασφάλειας στη συνεργασία. Πράγματι αυτή η προσέγγιση προς την ασφάλεια δεν είναι μοναχά το σήμα καθέν του ΟΑΣΕ. Είναι και το πιο, προ, πιο προωθημένη αντίληψη ασφάλειας σε ολόκληρο τον κόσμο γιατί είναι κάτι πολύ παραπάνω από απλή ισορροπία στρατιωτικών δυνάμεων και προϋποθέτει ότι οι αιτίε των κρίσεων, είτε πρόκειται για οικονομικές, είτε για ανθρωπιστικές, είτε για περιβαλλοντικές, πρέπει να αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα μαζί με τις στρατιωτικές μέσα σε διαφάνεια και σε ε, λήψη μέτρων αποκατάστασης εμπιστοσύνης. Στην βάση μιας ε, ασφάλειας μέσα σε συνεργασία. Με αυτό αυτό είναι που επαναζωογόνησαν οι χώρες μέλη με την πολιτική τους δήλωση του προηγούμενου Δεκεμβρίου ξαναδίνοντας ζωή στην διαδικασία αυτή από το Βανκούβερ μέχρι το Βραντιβοστόκ. Συνεχίζω κύριε Πρόεδρε. Στην, στις ίδιες ε, αρχές που βασίζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δηλαδή η ασφάλεια βασίζεται πρωτίστως στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν είναι συμπτωματικό λοιπόν ότι άρχισε η διαδικασία από μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζεται δραστήρια από όλες τις χώρες μέλη της Ένωσης σε ένα κοινό όραμα για την ασφάλεια της ε, Υπήρου μας σε συνεργασία με τους εταίρους μας. Και αυτά είναι θεμελιώδεις και αδιαπρομάτευτες αξίες. Αυτή είναι η απάντησή μας στις προκλήσεις ασφάλειας του 21ου αιώνα. Η Ελλάδα είναι υπερήφανη που είχε την ιστορική ευκαιρία να συμβάλλει με τον τρόπο αυτό από το 2009 και μετά αναβάνοντας την Προεδρία του ΟΑΣΕ. Uh, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση καταρχήν στην ακρόασή σας και για τη δυνατότητα που μου δίνεται να εκφράσω την άποψη της Ρωσίας στα πιο σημαντικά θέματα των διεθνών σχέσεων. Έχει μεγάλη σημασία το ότι ε, γίνεται η ακρόαση την 22 Ιουνίου, διότι μας υπενθυμίζει τη μεγαλύτερη εθνική τραγωδία στην σύγχρονη ιστορία της Ρωσίας καθώς και τον ηρωισμό του Σοβιετικού λαού που δεν μπορεί να απαξιωθεί δεν μπόρεσε να απαξιωθεί από τον ολοκληρωτισμό του Στάλιν. Τα εστιακά σημεία της παρουσίασής μου αφορούν την αρχιτεκτονική ευρωπαϊκή, της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Την χρειαζόμαστε. Δεύτερον, την πρωτοβουλία της Ρωσίας ποια είναι η ουσία της και τρίτον το μόνιμο ερώτημα για το τι μέλη γενέστε. Ήμουνα πρόσφατα στην διάσκεψη κορυφής Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένας Ευρωπαίος ανέφερε γιατί να αλλάξουμε το σύστημα, το υπάρχον σύστημα ασφάλειας εάν μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτό το σύστημα χωρίς τη Ρωσία. Μπορούμε να το επιτύχουμε χωρίς τη Ρωσία, όχι κατά της Ρωσίας βεβαίως. Και η αντίρρησή μου σε αυτό το σχόλιο, η απάντησή μου είναι διτή. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν μπορεί να ανατεθεί στην ευρωπαϊκή ε, Ένωση και το ΝΑΤΟ αποκλειστικά, διότι η απειλή έχει διεθνικό χαρακτήρα και γι' αυτό χρειάζεται η αρρωγή της Ρωσίας. Επειδή μοιραζόμαστε την Ήπειρο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ που διαθέτουν το μεγαλύτερο οικονομικό και στρατιωτικό δυναμικό. Χωρίς τη Ρωσία δεν θα μπορέσει να κινηθεί το ΝΑΤΟ, διότι η Ρωσία ήταν η ε, βασική δύναμη για τη διάλυση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και για τις ε, συνολικές διευθετήσεις ασφάλειας. Όλοι οι πόλεμοι τελείωσαν με συμφωνίες ειρήνης και συνολικής διευθέτησης θεμάτων ασφαλείας. Τίποτα δεν συνέβη με τη λήξη του ψυχρού πολέμου. Το γεγονός ότι η Ανατολή κατέρευσε δημιούργησε την άποψη στη Δύση ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα. Το προηγούμενο διτό ή διπολικό σύστημα ήταν βεβαίως πρωτόγονο αλλά διαδραμάτισε το ρόλο του. Ο ψυχρός πόλεμος έληξε πριν από 20 χρόνια, αλλά ανέκυψαν νέοι κίνδυνοι και απειλές. Εάν δούμε τη διάρθρωση ασφάλειας, βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με παλαιά θράψματα και με καινοτόμα στοιχεία τα οποία δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες. Μετά τον διπολισμό είχαμε την κρίση του Κωσυφοπεδίου το 1990 και την κρίση του Καυκάσου το 2008 που αποδεικνύουν ότι κανένα θεσμικό όργανο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις σειράξεις. Δηλαδή δεν αντιμετωπίστηκε η πρώτη μεταπολική, μεταδιπολική κρίση. Το ΝΑΤΟ και ο ΑΣΕ έχουν παραλύσει και το ΝΑΤΟ είναι μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης του προβλήματος. Μιλάμε για ε, γεωπολιτική επέκταση προς Ανατολάς και αυτή είναι η βασική πηγή του σκέλους της ασφάλειας ως προς τις σχέσεις ε, Μόσχας με τη Δύση. Όπως είπε και ένας Γερμανός συνάδελφος, το ΝΑΤΟ είναι η διπολική ιδέα στο μεταδιπολικό πλαίσιο, ιστορικό πλαίσιο. Και παράλληλα Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να είναι κανείς διαμεσολαβητής μεταξύ ΙΠΑ και Ρωσίας. Αλλά αυτό το επέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει στρατιωτικό χαρακτήρα. Ως προς την πρωτοβουλία Medvedev μπορώ να πω ότι το σοκ μετά την σύραξη του Καυκάσου οδήγησε σε συζητήσεις γύρω από την πρωτοβουλία Μετβέτεφ για μία νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας. Στην αρχή υπήρξε μεγάλος σκεπτικισμός από πολλούς ε, πολιτικούς αναλυτές και πολιτικούς που είπαν «Α, είναι κάτι παρόμοιο με την ε, πρωτοβουλία Γκορμπατσόφ για τον κοινό ευρωπαϊκό οίκο, Άλλοι είπαν ότι η πρωτοβουλία ΜΕΤΒΕΤΕΦ αποτελούσε στην ουσία μία σφήνα μεταξύ των συμφερόντων των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η πρωτοβουλία Μετβέντεφ θα πρέπει να ειδωθεί ως ένα μήνυμα ότι δηλαδή το υπάρχον αρχιτεκτόνιμα ασφάλειας δεν ήταν λειτουργικό, ήταν παροχημένο. Γι' αυτό και χρειαζόταν αναθεώρηση, πλήρης αναθεώρηση. Ένα χρόνο μετά η πρωτοβουλία οδήγησε στο προσχέδιο της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ασφάλειας. Ξέρετε βεβαίως την ουσία του κειμένου, γι' αυτό δεν θα ήθελα να την επαναλάβω, γιατί τρέχει και ο χρόνος. Απλώς θα μιλήσω για ορισμένα στοιχεία της συνθήκης που θα πρέπει να είναι δεσμευτική για όλες τις περιφέρειες από το Βανκούβερ μέχρι το ε, Βλαδιβοστόκ και επίσης αναφέρεται τις θέματα ασφαλείας όπως και στο Βορειοατλαντικό ε, Σύμφωνο. Βεβαίως, οι δυτικοί σύμμαχοι της Ρωσίας είπαν ότι δεν υπάρχουν οι βάσεις για μια δεσμευτική συνθήκη, διότι δεν υπάρχουν μηχανισμοί υποχρεωτικής εφαρμογής. Μιλάμε δηλαδή για σκληρή ασφάλεια όταν απειλείται η ευρωπαϊκή ασφάλεια γενικότερα. Αυτό ελέγχθη για αυτή τη σφήνα της Ρωσίας μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποια και να είναι όμως τα νομικά ερίσματα αυτής της πρότασης αντικατοπτρίζει δύο πραγματικότητες. Πρώτον, η σκληρή ασφάλεια έχει σημασία για τη Ρωσία και αν δεν υπάρχουν δραστικές αλλαγές θα αποτελέσει μείζον ζήτημα ενδεχόμενων απειλών με τη Δύση. Δεύτερον, ο δεσμευτικός χαρακτήρας που απαιτεί η Ρωσία απορρέει από την κακή της πείρα, από την εμπειρία δηλαδή που είχε με το ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα την επέκτασή του μετά την ενοποίηση της Γερμανίας. Βεβαίως, οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ δεν θα μπορούσαν να ζητήσουν την αρρωγή της ε, Ρωσίας για προστασία. Όμως αυτό είναι ένα στοιχείο που άπτεται άμεσα της ε, γενικότερης αμυντικής αρρωγής και θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα στοιχείο για έναν ευρύτερο ευρωπαϊκό διάλογο ασφαλείας για να αναθεωρήσουμε τις πολιτικές του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Ως προς την ε, παρέμβαση αυτή της Ρωσίας θα ήθελα να πω ότι δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχαν θεμελιώδη ζητήματα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Και το παράδοξο είναι ότι η κυβέρνηση Ομπάμα τόνισε το εύρος αυτών των βασικών διαφορών, διότι πλέον δεν είναι δυνατόν να κατηγορήσουμε την κυβέρνηση Μπούς. Δεν υφίσταται πλέον. Γνωρίζετε ότι και η Ρωσία και η Δύση αποφάσισαν να μην δημιουργήσουν νέους θεσμούς ούτε να καταρρύψουν τους ε, υπάρχοντες ούτε να διαλύσουν τους υπάρχοντες θεσμούς. Η ιδεατή λύση αφορά την επανακατανομή των παλαιών λειτουργικών και ρόλων της διάρθρωσης αυτής. Η οικονομική ασφάλεια αφορά τη συνεργασία της Τουρκίας, της Ουκρανίας, της Ρωσίας και της ε, κοινοπολιτείας ανεξαρτήτων κρατών, έτσι ώστε να ε, διασφαλιστεί ο ε, ανεφοδιασμός ενέργειας. Επίσης, ως προς την επίλυση διαφορών και την απαλυφή των εξτρεμιστικών κινημάτων, αυτό ακριβώς το σκέλος μπορεί να επιτευχθεί με τη συνεργασία της Ρωσίας. Μπορούν να ανακύψουν και διάφοροι μηχανισμοί και οργανώσεις διαμεσολάβησης. Το UCIS είναι ένα μέσον καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Η εξωτερική ασφάλεια της Ευρώπης, η απαλυφή των όπλων μαζικής καταστροφής, η μαζική πειρατεία μπορεί να παταχθεί με τη βοήθεια της ε, Ρωσίας, ιδιαίτερα ως προς την οργάνωση του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας, του CSTO, ως προς τα ανθρωπιστικά ζητήματα, εκπαίδευση, θεωρήσεις, όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν μέσω συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ΟΑΣΕ. Μετά την ε, συνθήκη της ε, Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας βασικός παίχτης για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και η ευρωπαϊκή ασφάλεια αποκτά ολοένα και ευρύτερο ρόλο. Ο μελλοντικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς σχέσεις θα βασιστεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και στην οικοδόμηση νέων εταιρικών σχέσεων πέρα από τις ε, δομές της. Γιατί η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος και ο κυριότερος γείτονάς της. Ως προς το ΝΑΤΟ θα πρέπει να ασχοληθεί με το ευρωατλαντικό σκέλος καθαρά και να τεθούν ε, νέα πλαίσια για την για τον μεταδιπολικό ατλαντισμό. Ο κύριος Μπουτικόφερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι απευθεία, στα όσα είπε η κυρία Αρμπάτοβα. Είπατε ότι χωρίς τη Ρωσία σημαίνει ενάντια στη Ρωσία. Δεν ξέρω αν μας βοηθεί αυτή η διαδική λογική. Κανένας από εμά δεν λέει χωρίς τη Ρωσία. Με τη Ρωσία βέβαια δεν μπορεί και να σημαίνει σύμφωνα με ρωσικές συνταγές. Ευχαριστώ την κυρία Αρμπάτοβα που ξεκαθάρισε τόσο καλά ότι στην βάση της πρωτοβουλίας, στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας που αναπτύξατε, φαίνεται πως υπάρχει ιδέα ότι το ΝΑΤΟ είναι το βασικό πρόβλημα. Αυτό διευκρινίζει λίγο τα πράγματα. Τώρα, έχω μια ερώτηση για τον κύριο Σιλβέστρη. Αν κατανόησα καλά, είπατε κύριε Σιλβέστρη ότι καθήκον, το καθήκον του ΝΑΤΟ να διοργανώνει τη συλλογική άμυνα είναι, εάν το πάρει κανεί αυστηρά, όλο, ε, αμφισβητείται μάλλον όλο και περισσότερο. Διότι με τη στρατηγική των συνασπισμών των προθήμων υπονομεύεται η αλληλεγγύη αυτή. Αν καλά το κατάλαβα, αν αυτή είναι η ανάλυση σας, διαρωτώ με τότε που εντοπίζετε εσείς τότε το ποιο είναι το καθήκον της συλλογική άμυνας ή καθίσατε πλέον περίτη αυτή. Και μία ερώτηση για τον κύριο Χάμιλτον. Αφού πρώτα πω ότι χαίρομαι για το ότι αναγνωρίζετε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα από τους τρεις πυλώνες και πράγματι οι πυλώνες αυτοί συχνά εμποδίζουν ένα τον άλλο. Τώρα από αυτό έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτο, ίσως και να μην άκουσα βέβαια καλά. Η Ένωση ως ένας από τους τρεις ευρωπαϊκούς πυλώνες έχει κάποιο ρόλο να παίξει και στον χώρο home security. Παίζουμε τον ρόλο αυτό με την Αταλάντη για παράδειγμα. Μα συγγνώμη, διορθώνει ο, ο διερμηνέας, όχι home security αλλά hard security, την σκληρή ασφάλεια. Λοιπόν, υπάρχει εδώ ένας ρόλος να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο, εάν γίνει κατανομή έργου μεταξύ των διαφόρων θεσμών, παραμένει ωστόσο το θέμα της ολοκλήρωση όλων αυτών των συμβολών, α το πω έτσι. Πώ συντονίζεται αυτό. Εγώ βλέπω να διαμορφώνεται μέσα από αυτά που ε, λέει η ομάδα της κυρίας Όλμπραϊτ βλέπω να υπάρχει μια κίνηση προς μια ευρωπαϊκοποίηση του ΝΑΤΟ. Μήπως πρόκειται δηλαδή για επικάλυψη, ότι δηλαδή ναι μεν δεν προχωρούμε σε κατανομή έργου, αλλά από την άλλη μεριά θεωρούμε ότι το ΝΑΤΟ είναι αρμόδιο για τα πάντα. Τρίτο, ο ρόλος της πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Ουάσιγκτον δέχομαι διαφορετικά μηνύματα. διαβάζοντας για παράδειγμα τα όσα λέει ο Τζοε Μπάιντεν στην International Herald Tribune η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί στο άρθρο που λέει το μέλλον της Ευρωπαϊκής ε, Υπήρου δεν αναφέρει καθόλου την Ευρωπαϊκή Ένωση άλλα λέει αυτός άλλα λέει ο Χίλαρη Κλίντον η Χίλαρη Κλίντον είπε αυτά που είπε ο Μπάιντεν στο Παρίσι ή χρειάζεται εν πάση κάποια στιγμή να καθίσει η Αμερικανική κυβέρνηση και να αποφασίσει τι θέλει. Λαντσμπέργκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι ερωτήσεις μου αφορούν κυρίως τους κυρίους Σιλφέστρη και Χάλμιλτον. Όπως θυμάμαι από την προηγούμενη μου ζωή, ο πρόεδρος Γέλσιν το 1993 είχε την ιδέα για μια ευρωπαϊκή συνθήκη ασφαλείας που θα αντικαθιστούσε το ΝΑΤΟ ως παροχημένο, όπως παροχημένη ήταν και η συνθήκη, το σύμφωνο της Βαρσοβίας προκειμένου να υπάρξει μια κοινότητα και με τη Ρωσία και έτσι θα είχαμε μια νέα πολιτική ατζέντα για την Ευρώπη όπου τίποτα δεν θα γινόταν χωρίς την Ρωσία. Και ενδεχομένως θα μπορούσαμε να έχουμε μια κοινή ήπειρο της Ευρώπης διαχωρισμένη από τους υπόλοιπους του Ατλαντικού. Βεβαίως, εμείς δεν ήμασταν τόσο αφελείς. Και αυτό μας επέτρεψε να σώσουμε τα Βαλκάνια. Η έννοια λοιπόν του ότι τίποτα χωρίς τη Ρωσία φαίνεται να επανέρχεται σήμερα. Και μας λέτε ότι ό,τι και να κάνουμε χωρίς τη Ρωσία παρανοϊκά η Ρωσία θα το ερμηνεύει ως κατά της Ρωσίας. Υπάρχουν περιοχές όπως το Καραμπάχα που δεν μπόρεσαν να την καταλάβει η Αρμενία χωρίς τη Ρωσία. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουμε δηλαδή δράση χωρίς τη Ρωσία. Και αναρωτιέμαι, αυτή η νέα πρόταση Μετβέντεφ προσθέτει κάτι με βάση και τα παραδείγματα στον Κάφκασο ή αποτελεί απλό αντίγραφο ενός παλιού αριστοργήματος. Και αν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές με το παρελθόν, ποιες είναι σε αυτές. Ευχαριστώ. Δύο άτομα έχουν ζητήσει το λόγο που είχαν ζητήσει και πριν το λόγο. Η κυρία Λέζιν και η κυρία Γκόμες. Σας παρακαλώ να ξεχάσετε τις ερωτήσεις και απλά να απαντήσουν οι ομιλητές στις ερωτήσεις που μόλις έγιναν. Γιατί έχουμε ένα ακόμη πολύ σημαντικό θέμα να συζητήσουμε και μόλις κατέφτασε και ο κύριος Μπροκ που θα μας το παρουσιάσει. Σας παρακαλώ λοιπόν να μου το επιτρέψετε αυτό. Θα δώσω τώρα το λόγο στους ομιλητές για να απαντήσουν και θα κλείσουμε εδώ τη συζήτηση για να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Εκτός μικροφώνου η παρατήρηση της κυρίας Κόμες. 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε κυρία Γκόμες. Κυρία Λέσσιν, 30 δευτερόλεπτα, αν θέλετε. Κυρία Γκόμες. Συμφωνείτε κυρία Μαρινάκη με τον κύριο Χάμιλτον ότι η αποστολή στη γεωργία του ΟΑΣΕ θα μπορούσε να επιτελέσει αυτή την εργασία σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Μπατόβα η οποία διαφωνεί θεωρεί ότι ο ΑΣΕ είχε, ήταν ανενεργός και προς την κυρία Νάντια Μπατόβα, πιστεύετε ότι αυτή η επιφυλακτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπει σε ένα νέο αρχιτεκτόνιμα ασφαλείας μαζί με τη Ρωσία σχετίζεται με το γεγονός ότι υπάρχει καχυποψία για το κατά πόσο η Ρωσία είναι μια δημοκρατική δύναμη και έχει κατασταλτικούς τρόπους αντιμετώπισης θεμάτων όπως στην Τσετσενία, στον Κάφκασο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είπατε τίποτα χωρίς τη Ρωσία. Μήπως όμως είναι προβληματικό το ότι στην στρατηγική του ΝΑΤΟ 2020 λέει αναφέρεται η φιλική σχέση με την Ρωσία, από την άλλη μεριά όμως τονίζεται ταυτόχρονα και το ενδεχόμενο η Ρωσία να κινηθεί προς μια εχθρική κατεύθυνση. Μήπως αυτό όμως γίνεται μια αυτοεπαληθευόμενη προφητεία και ένα σύστημα ασφάλειας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα θεμητά συμφέροντα όλων των συμμετεχόντων. Νομίζω ότι το ΝΑΤΟ 2020 δεν το πράττει αυτό. Εξακολουθεί να υπάρχει η πολιτική της ανοιχτής πόρτας, κυρίως ό,τι αφορά Γεωργία και Ουκρανία. Θα παρακεστώ σε αυτά και αναμένω την απάντησή σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σιλβέστρη, καταρχάς και Χάμιλτον και μετά Μαρινάκη και Αρμπάτοβα. Για τον κύριο Μπούτικοφ να πω ότι είπα ότι το ΝΑΤΟ προσφέρει λιγότερη ασφάλεια σήμερα από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν άλλα θεσμικά όργανα που μπορούν να προσφέρουν συλλογική άμυνα. Απλά αυτή τη στιγμή έχουμε μείωση της συλλογικής άμυνας. Η βασική προϋπόθεση, η βασική μας ανάγκη στην Ευρώπη, αν θεωρούμε ότι δημιουργείται μια νέα απειλή που θα απαιτήσει συλλογική άμυνα, η μόνη μας ανάγκη τότε θα είναι να έχουμε τη ΣΥΠΑ στην στο πλευρό μας για να στηρίξουν τις ανεπαρκείς δυνάμεις μας. Το πρόβλημα βεβαίως είναι να διασφαλίσουμε ότι θα είναι κοντά μας οι Ηνωμένε Πολιτείε όταν θα τις χρειαζόμαστε. Και αυτό σήμερα δεν είναι τόσο σίγουρο όσο στο παρελθόν. Ας το πούμε ως εξή. Δεν νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να καταστρέψουν το ΝΑΤΟ. Μόνο οι Ηνωμένε Πολιτείε μπορούν να καταστράψουν το ΝΑΤΟ. Όχι να το καταστρέψουν, αλλά να μειώσουν το ρόλο του, γιατί το ΝΑΤΟ δεν θα μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες που ζητούν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε όχι τόσο για την αλλαγή ή την μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ αλλά για την καλύτερη κατανόηση Ευρωπαίων και Αμερικανών. Και εδώ η Ευρώπη καλύτερα θα ήταν να εκπροσωπηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ρωτήσουμε τους Αμερικανούς τι θέλουν να επιτύχουν για το μέλλον τους. Τώρα, το ερώτημα που ετέθη για τον Γέλσιν το 1993 Δεν ξέρω τι θα πούν η κυρία Αρμπάτοβα και οι υπόλοιποι, αλλά να πω ότι φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ για την Ρωσία και για το κατά πόσο μπορεί να καταλάβει η Ρωσία περί τίνος πρόκειτο. Βλέποντας το έγγραφο για την στρατιωτική στρατηγική της Ρωσίας, θεωρώ ότι ουσιαστικά το Υπουργείο Αμήνης και το Γενικό Επιτελείο της Ρωσίας εξακολουθούν να θεωρούν ότι η βασική απειλή για τη Ρωσία είναι το ΝΑΤΟ. Και επίσης κάνουν και μία διάκριση μεταξύ των κύριων απειλών και των κινδύνων που πρέπει να τους, ε, να υποστούν. Είναι λοιπόν δύσκολο να καταλήξουμε σε ένα κοινό έγγραφο ασφαλείας αν θεωρείται το ΝΑΤΟ βασική απειλή. Εγώ δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να φοβόμαστε μία κυριαρχία ρωσική στην Ευρώπη ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αντίθετο μάλλον ισχύει. Οι Ρώσοι φοβούνται μία οικονομική και πολιτιστική επικυριαρχία της Δύσης στη Ρωσία. Όμως είναι γεγονός ότι δεν έχουμε έναν σαφή ορισμό των Ρώσων για το τι εστί η ασφάλειά τους και αυτό το χρειαζόμαστε. Ο κύριος Κόφερ μου έθεσε ορισμένα ερωτήματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως προς την εξωτερική ασφάλεια θα ήθελα να πω ότι τα Βακάνια, δεν ξέρω κατά πόσο μιλάμε για σκληρή ε, ασφάλεια, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ετέθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το υποστήριξε η ΕΠΑ. Δηλαδή, η ΕΠΑ το ανέθεσαν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας τομέας λοιπόν όπου η ΕΠΑ ε, υποστήριξαν τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα σκληρής ασφάλειας. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με θέματα δόγματος, αλλά έχουμε να κάνουμε με τις ίδιες δυνάμεις που στέκονται σε διάφορα θεσμικά όργανα και δεν συνομιλούν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι θέμα ΝΑΤΟ κατά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τι θέλουμε να κάνουμε μαζί και τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις, ε, τους κινδύνους ασφαλείας μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Τη δεκαετία του 90 θεωρούσαμε ότι κάποιος φορέας πρέπει να κινηθεί πρώτος. Πρώτα το ΝΑΤΟ ή πρώτα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα νομίζω ότι αρκούμεθα με τις δυνάμεις μας. Άρα αυτή η παλαιά συζήτηση δεν έχει νόημα. Έχουμε το, τη συμφωνία Βερολίνο ΣΥΝ, Berlin ΠΛΑΣ» για να δούμε κατά πόσο το ΝΑΤΟ μπορεί να βοηθήσει και τη ΣΥΠΑ σε ορισμένες περιπτώσεις. Μιλάμε δηλαδή για σκληρή ασφάλεια όπως στην περίπτωση του Κονγκό. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αναλάβει αυτές τις αποστολές. Εμείς θα πρέπει να προστρέξουμε και να σας ε, βοηθήσουμε με τα ε, αεροπορικά μας μέσα. Άρα θα πρέπει να αποφασίσετε το ΝΑΤΟ θα το κάνει αυτό ή δεν θα το κάνει. Θα το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας όμως πρόσβαση στον εξοπλισμό του ΝΑΤΟ. Ή και οι δύο φορείς θα κινηθούν στα Βαλκάνια, στο Αφγανιστάν και πάλι φτάνουμε στην Συμμαχία των Προθήμων. θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θέλουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις προκλήσεις ασφάλειας. Μπορούμε να βρούμε το αντίστροφο Berlin Plus, διότι το ΝΑΤΟ δεν κάνει πολλά πράγματα στο πολιτικό τομέα που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα χρειαζόμαστε τα δικά σας εφόδια ως προς το μη στρατιωτικό σκέλος. Αυτή είναι μια θεμητή συζήτηση. Το τελευταίο σας ερώτημα Ω ως προς την αμφιθυμία των ΗΠΑ ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η, η Εξ Κλίντον ήταν απόλυτα σαφή στο Μάρτιο. Είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει ε, κάποια προθυμία ως προς συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Μιλάμε και για ένα μη στρατιωτικό πυρήνα και ο πρέσβης μας έχει έρθει στις Βρυξέλλες πολλές φορές για να δούμε πώς θα συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανταποκρίθηκε πολλές φορές. Ξέρουμε, έχουμε καταλόγους χωρών που βρίσκονται σε κίνδυνο, αλλά δεν συμμεριζόμαστε, δεν μοιραζόμαστε αυτούς τους καταλόγους, αυτά τα δεδομένα. Γιατί να μην γίνει ανταλλαγή προσωπικού ως προς το πολιτικό σκέλος, δηλαδή το μη στρατιωτικό, όπως ζητήσαμε από την κυρία Άστον. Εσείς έχετε απορρίψει αυτές τις ε, προτάσεις, άρα δεν μπορείτε να πείτε ότι οι ΙΠΑ δεν έχουν προσπαθήσει. Αλλά υπάρχει αυτή η αμφιθυμία των ΙΠΑ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντικατοπτύσσει την αμφιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον ίδιο το, το ίδιο της το θεσμικό πλαίσιο. Και η συνθήκη της Λισαβόνας είναι ένα πολύ πρόσφορο παράδειγμα. Στην Ουάσιγκτον θεωρούμε ότι επιδεινώθηκαν τα πράγματα για το πώς θα συνεργαστούμε, διότι είναι συγκεχημένη εικόνα από τότε που εγκρίθηκε η συνθήκη της Λισαβόνας, ενώ για οκτώ χρόνια μας λέγατε ότι υπάρχει ένας τηλεφωνικός αριθμός για να επικοινωνούμε μαζί σας. Εμείς δεν κατανοούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν βρισκόμαστε εδώ. Είναι η πιο σημαντική οργάνωση στον κόσμο στην οποία δεν ανήκουμε, όπως πάντα λέω, αλλά θα πρέπει να την κατανομήσουμε. Και νομίζω ότι εκεί έγκυται η αμφιθυμία των ΗΠΑ, ότι δεν κατανοούμε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Μαρινάκη έχει το λόγο και η κυρία Αρμπάτοβα στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Εκ των υστέρων, ακόμη και η υπέρμαχοι της διακοπής λυπούνται που δεν παραμένει η Προεδρία και προσπαθούν να την... Ναι, η παρουσία με συγχωρείτε μάλλον και προσπαθούν να έχουν και τέτοια να αποκτήσουν παρουσία στην Γεωργία προκειμένου να υπάρχει και κάποιος άλλος μάρτυρας για το τι συμβαίνει επί τόπου όσον αφορά τις δραστηριότητες των δύο πλευρών και επίσης να πω ότι δημιουργήθηκε μία μαύρη τρύπα στο θέμα της ε, δημιουργίας δημοκρατικών θεσμών στη Γεωργία. Και αυτό ήταν βασική δραστηριότητα του ΟΑΣΕ και κανένας δεν μπόρεσε να αναλάβει αυτό το ρόλο. Γενικά λοιπόν πήραμε τα διδάγματά μας. Βεβαίως όταν κάτι πεθάνει είναι δύσκολο να το αναβιώσουμε. Και εμείς θεωρούμε ότι είχαμε ένα πτώμα στο νεκροτομείο για έξι μήνες και δεν εγκαταλείπαμε παρόλα αυτά, αλλά τελικά 30 Ιουνίου αποφασίσαμε να καταλάβουμε πώς έχει η κατάσταση, εγκαταλείψαμε, αλλά ελπίζουμε παρόλα αυτά ότι θα είναι καλύτερη η συνέχεια στο μέλλον. Κύριε Αρπάτοβα, κάποια πράγματα για τον ΝΑΤΟ να διορθώσω λίγο τον Στέφανο. Στο στρατιωτικό δόγμα του ΝΑΤΟ η επέκταση αναφέρεται ως κίνδυνος, όχι ως απειλή. Και αναφέρεται συγκεκριμένα η επέκταση των στρατιωτικών υποδομών του ΝΑΤΟ κοντά στα σύνορα της Ρωσίας. Αν στο τέλος ε, της διπολικότητας το ΝΑΤΟ είχε ολοκληρώσει τις εσωτερικές του μεταρρυθμίσεις και είχε βρει μια νέα ταυτότητα, δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα. Δεν μπορούμε να είμαστε δύο σε ένα και στρατιωτική συμμαχία και ασφάλι, θεσμός ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να είμαστε ο λίγον τι έγκυοι. Όσον αφορά τώρα τις τοπικές κρίσεις, οφείλονταν σε τοπικούς παράγοντες. Όμως, καταλαβαίνετε νομίζω ότι ο βασικός λόγος ήταν η σχέση Ρωσίας και ΝΑΤΟ και οι ανησυχίες της Ρωσίας κρίση στον Κάφκασο είχε να κάνει με τις σχέσεις Ρωσία και ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα όσον αφορά τον ΟΑΣΕ. Η Ρωσία ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης μετά, μετά τον τέλος του ψυχρού πολέμου για τον ρόλο του ΟΑΣΕ. Όμως δυστυχώς η Δύση δεν ενδιαφερόταν καθόλου για το μετασχηματισμό του ΟΑΣΕ. Μετά τον ψυχρό πόλεμο είχαμε δύο οργανισμούς ασφαλείας. Το ΝΑΤΟ για τις εξωτερικές περιοχές και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΑΣΕ για την κοινοπολιτεία ανεξαρτητών κρατών. Παρόλα αυτά, αν και συνειδητοποιούμε ότι παραμένει βασικό φόρουμ. Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος ο ΑΣΕ είναι αυτός που αποφάσισε να μετατοπιστεί προς το γεωγραφικό χώρο ανατολικά της Βιέννης και προς θέματα ανθρωπιστικά. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει μετασχηματισμός του ΟΑΣΕ σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τέλος του διπολισμού. Τώρα όσον αφορά τις σχέσεις Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, σίγουρα υπάρχει βαθιά δυσπιστία μεταξύ των δύο. Γιατί με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, νομίζω και από τις δύο πλευρές οι προσδοκίες ήταν υπερβολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ήλπιζε ότι η Ρωσία θα γίνει μια ευημερούσα δημοκρατία μέσα σε μια νύχτα. Η Ρωσία ανέμενε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή μετά το τέλος του διπολισμού. Και αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε γιατί παρόλο που αρκετοί θεωρούν τη δεκαετία του 90 ως την καλύτερη περίοδος της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, τότε ελήφθη η απόφαση για επέκταση του ΝΑΤΟ, η οποία μετά έγινε και η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτό που είδαμε ήταν ότι η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ στην μετακομμουνιστική Ευρώπη έγινε βασική προϋπόθεση, απαραίτητη προϋπόθεση για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα δηλαδή ένταξη στο ΝΑΤΟ, μετά προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λοιπόν το ΝΑΤΟ έπαιξε πολύ αρνητικό ρόλο. Όμως μια εταιρική σχέση για εξυγχρονισμό θα μπορούσε να θέσει τις σχέσεις μας σε νέες βάσεις γιατί ο οικονομικός εξυγχρονισμός πρέπει να συμβαδίζει με το πολιτικό εξυγχρονισμό. Αν θέλουμε να αυξήσουμε τις ξένες επενδύσεις, πρέπει να έχουμε το κατάλληλο εγχώριο περιβάλλον για τους επενδυτές. Άρα η Ρωσία βαθμιαία θα εκδημοκρατιστεί. Ευχαριστώ. Κύριος Λίσακ, να συνοψίσει. Θα είμαι σύντομος, άλλωστε υποσχέθηκα. Πρώτα πρώτα βλέπω τους κυρίους Μπροκ και Σάριους Βόλσκι που θέλουν να μιλήσουν για την υπηρεσία εξωτερικής δράσεως. Δεν φταίμε εμείς, δεν φταίμε εμείς. Αυτό θέλω να πω γιατί η συζήτησή μας άρχισε με καθυστέρηση. Άκουσα ορισμένους να μιλούν για την έκθεση της ομάδας της κυρίας Όλμπραϊτ. Δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα. Κάτι τέτοιο είναι mission impossible ισχυρίζονται ορισμένοι ότι θα τα λύσει όλα. Δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Είναι η αρχή τη συζήτηση. Εμεί θα πρέπει να συνεχίσουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει την συζήτηση με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και μελών βέβαια των Εθνικών Βουλών. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να πω ευχαριστώ στους ομιλητές και εμπειρογνώμονες. Είμαι βέβαιος ότι δεν είναι η τελευταία συζήτηση αυτή που κάναμε μαζί σας. Uh, uh, σας ευχαριστούμε όλους και τους ε, προσκαλεσμένους μας και τώρα περνάμε στο τελευταίο θέμα της ε, σημερινής ε, ημερήσιας διάταξης που είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και θα ήθελα να σας πω ότι στις 21 Ιουνίου τη Δευτέρα στη Μαδρίτη ο κύριος Μπροκ μαζί με τους Φερχόφστατ και Γκουαλτιέρη συμμετείχαν σε μία συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με την Προεδρία του Συμβουλίου και με την ύπατη εκπρόσωπο για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Φτάσαμε λοιπόν σε μία απόφαση για την σύσταση της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θα ήθελα ο κύριος Μπρόκ να μας κάνει μια παρουσίαση των αποτελεσμάτων και μετά θα γίνει συζήτηση. Ο κύριος Μπρόκ, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλήξαμε σε μια συμφωνία που δεν μας δεσμεύει στην νομοθετική διαδικασία, θα ακολουθηθεί η συνήθις διαδικασία. Αυτό περιλαμβάνεται και στην δήλωση των συμμετεχόντων ότι ο καθένας δηλαδή θα επιζητήσει υποστήριξη εντός του θεσμικού του οργάνου και εν προκειμένου η Επιτροπή Εξωτερικών είναι η αρμόδια επί της ουσίας στην Ευρωβουλή. Τις, τις επόμενες ημέρες θα αποφασίσουμε πώς θα κινηθεί περαιτέρω η διαδικασία. Για μένα είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε στη συνήθεια διαδικασία τα καταστατικά του προσωπικού και τα λοιπά πριν από τις θερινές διακοπές. Η πορεία θα εξαρτηθεί πολύ και από το τι θα αποφασίσουν οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων. Αύριο το πρωί θα συναντηθεί ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου με τους επικεφαλής με τους πρόεδρους δηλαδή, των κοινοβουλευτικών, ε, με των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ο κ. Γκουαλτιέρη έπαιξε επίση σημαντικό ρόλο και θεωρεί ότι σε πολλούς τομείς έχουμε προχωρήσει και πολύ μάλιστα και ότι θα ήταν ίσως σκόπιμο να οι δεσμεύσει και να ολοκληρωθούν τμήματα τη διαδικασίας ώστε να μην υπάρξει αργότερα η δυνατότητα ορισμένη να αποχωρήσουν εντός εισαγωγικών, να υπαναχωρήσουν καλύτερα από την συμφωνία αυτή. Αυτά θα τα υποβάλω εγώ αύριο στο σχέδιο εκθέσεώ μου. Που θα έχει το ίδιο περιεχόμενο με αυτήν του κυρίου Φερχόφστατ. Ώστε να μην χρειάζεται να κάνουμε περαιτέρω δουλειά. Θα δούμε μετά πότε είναι η προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών. Ακούω ότι η Συνταγματική Επιτροπή αποφάσισε να βάλει την Δευτέρα λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών, μετά να συζητηθεί στις ε, πολιτικές ομάδες και την παραπάνω Δευτέρα πλέον στο Στρασβούργο να το συζητήσει στις 6 ώρα το απόγευμα, εμείς στις 9 το βράδυ δηλαδή, με τη συνεργασία του Σίλβιου Κονσάτο να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε κάποια ώρα να συζητήσουμε την Τρίτη το πρωί. Εάν την Πέμπτη θα καταλήξουμε σε απόφαση της Ολομέλειας, αυτό θα το δούμε ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν. Πάντως να έχουμε τη δυνατότητα να το πράξουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι ο καλύτερος δρόμος. Θα σας υποβάλω μια πρόταση που ανταποκρίνεται ακριβώς στο αποτέλεσμα των χθεσινών συζητήσεων. Όποιος δεν συμφωνεί μπορεί να κάνει τροπολογίες. Και αν οι τροπολογίες αυτές υποστηριχθούν από τόσους ώστε να τροποποιηθεί το περιεχόμενο της ε, έκθεσης, τότε θα θεωρήσω ότι εμείς οι τρεις διαπραγματευτήκαμε εσφαλμένα. Ελπίζω πάντως και σήμερα και τις επόμενες ημέρες και στις συνεδριάσεις που θα γίνουν εδώ αλλά και σε επιμέρους συνομιλίες όσων επιθυμούν θα μπορέσω να κερδίσω την υποστήριξή σας. Θέλαμε να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική υπηρεσία. Δική μας επινόηση άλλωστε ήταν η υπηρεσία εξωτερικής δράσης μέσα στην συνέλευση που προετοίμασε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θέλαμε, θέλαμε επίσης να μιλούμε με μία φωνή μέσα στην παγκόσμια τάξη. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης και η ύπατη εκπρόσωπος είναι υβριδικά όντα και έχουν αφενός κοινοτικές αρμοδιότητες και αφετέρου διακυβερνητικές. Και όλα αυτά είναι εξαιρέσεις της αρμοδιότητας της ΚΕΠΑ. Και γι' αυτό έχει και εντολή η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος να συντονίζει και να καθιστά δυνατή την ενότητα των εξωτερικών σχέσεων και διευθύνει την εξωτερική πολιτική. Έχει μόνο συντονιστικό ρόλο. Για να διασφαλίσουμε την κοινοτική μέθοδο και παραπέμπουμε και στην συνθήκη. Για τις πιο σημαντικές πολιτικές όπως την πολιτική αναπτύξεως, πολιτική γειτονίας, η είπατε εκπρόσωπος συντονίζει, οι υπηρεσίες συνεργάζονται, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εξωτερικής δράσεως. Η είπατε εκπρόσωπος μαζί με τον αρμόδιο επίτροπο υποβάλλει προτάσεις για την ελήψη αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την ευθύνη των Επιτρόπων Αναπτύξεως ή Γειτονίας. Όλα τα επιχειρησιακά μέσα που έχει στη διαθεσή της είπατε εκπρόσωπος περιλαμβάνονται στο τμήμα 3 επομένως και οι πόροι της ΚΕΠΑ εντασσόμενα έτσι στις κοινοτικές αρμοδιότητες και άρα και στα δικαιώματα του Κοινοβουλίου για τον δημοσιονομικό έλεγχο και τη χορήγηση απαλλαγής. Εμείς θελήσαμε αυτή η υπηρεσία να ενταχθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τον επιχειρησιακό της προϋπολογισμό λοιπόν υπάρχει ένα τμήμα 10 μόνο για τον επιχειρησιακό της προϋπολογισμό όπου διευκρινίζεται και λέμε και σε πολλά επιμέρους στην πράξη τμήματα και ο κύριος Γκουαλτιέρη που είναι πιο αρμόδιος μπορεί να σας πει λεπτομέρειες καλά ορισμένα τα γνωρίζω κι εγώ ότι πρέπει να δούμε δηλαδή ότι εδώ οι κανόνες εφαρμόζονται πλήρως οι κανόνες που ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ε, προπολογισμό, τον έλεγχο του προπολογισμού και την απαλλαγή. Τώρα πριν να ληφθούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου, όλες οι αποφάσεις και οι στατιωτικές πάνε στην υπηρεσία εξωτερικών δράσεων και δεν ισχύει πλέον η Συμφωνία Κυρίων που ίσχυε μέχρι τώρα όταν τα θέματα αυτά εντάσσονται σε αρμοδιότητες του Συμβουλίου Υπουργών. Επομένως, περιλάβαμε ορισμένα πράγματα ακόμα στην κοινοτική αρμοδιότητα. Και ε, δείτε και την υπόθεση της accountability, την οποία συζητήσαμε ήδη στην τελευταία συνεδρίαση. Λέει ότι και στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, στο μέλλον, η ύπατη εκπρόσωπος, οι, οι εκπρόσωποι της, έρχονται και αναφέρουν στην Επιτροπή Εξωτερικών πριν από την λήψη των αποφάσεων για εξωτερικές δράσεις αποφεύγουμε έτσι τα διάφορα με τους επιτρόπους κτλ. Και στα δύο έγγραφα, την statement δηλαδή της είπα της εκπροσώπου, αλλά και την πρόταση που θα βάλουμε στην Ολομέλεια, αυτά λέει η συμφωνία. Τα συντονίζουμε και με το πρακτικό, με το πρωτόκολλο μάλλον του Συμβουλίου, και αυτά δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα τη Ευρωπαϊκής Ένωση, ώστε να υπάρχει ένας ενίο χαρακτήρας. Και επειδή δημοσιεύει το Συμβούλιο, άρα δεν είναι μονάχα δεσμευτικέ δηλώσει αυτές που θα δημοσιεύονται τη είπα τη εκπροσώπου, αλλά και του Συμβουλίου. Αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία για την δεσμευτικότητα των αποφάσεων αυτών. Μετά υπάρχουν και διάφορες λεπτομέρειες του προϋπολογισμού των ελέγχων για να ικανοποιήσουμε και τους ε, βουλευτές της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού Για το προσωπικό τουλάχιστον ένα τρίτο του προσωπικού θα είναι εθνική αξιωματούχοι η οποία όμως εθνική αξιωματούχοι και αντίθετα με αυτό που ισχύει τώρα και που απαγορεύει. Μπορούν να υποβάλουν αιτήσει να προσληφθούν ως μόνιμοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διαγωνισμούς, βέβαια, στη βάση των προσόντων τους. Τους ανοίγουμε λοιπόν τη δυνατότητα να κάνουν σταδιοδρομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον υπάρχουν θέσεις και εφόσον έχουν τα σχετικά προσόντα, να μπουν στην εξωτερική υπηρεσία ώστε να τους να λύσουμε αυτήν την μονομερή πίστη υπακοή δηλαδή στις εθνικές αρχές και διοικήσεις. Είναι μια λεπτομέρεια που έχει όμως τεράστια σημασία. Επίσης, στο μέλλον τουλάχιστον 60% τουλάχιστον 60% όλων των υπαλλήλων θα πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν κάνουμε εδώ διάκριση μεταξύ Συμβουλίου και Κομισιόν. Μετά από μια μεταβατική περίοδο όπου θα διορίζονται ευθέως τα πρόσωπα αυτά, μετά θα, δεν θα προέρχονται πλέον από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή, από την Κομισιόν δηλαδή, αλλά θα προσλαμβάνονται ευθέως ως υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προσωπικό από τις χώρες μέλη θα χρησιμοποιείται πλέον μονάχα για ειδικέ αποστολές, για παράδειγμα και ένστολο προσωπικό. Και αυτό είναι ένα πρόσθετο μέτρο ασφάλειας. ώστε να αποφύγουμε οποιαδήποτε επιστροφή τώρα της ε, υπηρεσίας αυτής στο διακυβερνητικό επίπεδο, έστω και από το παράθυρο. Σημαντικός θα είναι ο ρόλος της παρούσας επιτροπής, όπως είπα, και για τους εκ των προτέρων ελέγχους στον τομέα της κοινή εξωτερικής και πολιτικής ασφάλειας, που είναι πολύ αρμοδιότερη η παρούσα επιτροπή, και σε ό,τι αφορά την, τον έλεγχο εμπιστευτικών εγγράφων. Μέχρι τώρα έχουμε αυτή την πενταμελή επιτροπή που μπορεί να δέχεται εμπιστευτικές πληροφορίες. Εμείς θα το διευρύνουμε αυτό και ορίζεται τώρα ότι όταν γράφει στην κυρία Άστον, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, η πρόεδρος της Επιτροπής για να επιτραπεί η πρόσβαση κάποιου ειδικού εισηγητού σε κάποια εμπιστευτικά έγγραφα. Αν πρόκειται για το Αφγανιστάν, για παράδειγμα, θα μπορεί τότε ο Μπούζεκ και ο Αλμπερτίνη να γράψει στην Άστον και να παρακαλέσει να επιτραπεί η πρόσβαση του Χ, του Υ ή του Ψ βουλευτού στην, ε, σε ε, ορισμένα εμπιστευτικά έγγραφα. Αυτό είναι σημαντικό. Εγώ ο ίδιος υπήρξα πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών τον προηγούμενο αιώνα βέβαια ήταν αυτό, και ήταν ένα από τα όνειρά μας να έχουμε αυτήν την απριόρι δυνατότητα εξέτασης των εμπιστευτικών εγγράφων. Και τώρα να, το πετυχαίνουμε. Και νομίζω ότι για την Επιτροπή Εξωτερικών πρόκειται για αποφασιστικής σημασίας βελτίωση της κατάστασης και για θέματα political accountability. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και απέναντι στις Εθνικές Βουλές. Άλλωστε και τα δικαιώματά μας για τον προπολογισμό, τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει κατάλληλα μαζί συνεργασία με τους βουλευτές της Επιτροπής Προπολογισμών. Τώρα ενισχύονται οι δυνατότητες αυτές, αυτά περιλαμβάνονται μέσα στην συμφωνία, ότι δηλαδή η ότι εκπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπείται από επιτρόπους για θέματα κοινοτικά ή και μεικτά και εφόσον νομιμοποιούνται επίσης εκπρόσωποι του Συμβουλίου και έχουμε τότε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε συζητήσεις εξωτερικής πολιτικής και στις, και στις ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές και στην Ολομέλεια, για παράδειγμα για θέματα πυρηνικών εξοπλισμών, ή για παράδειγμα για την Ινδία, θα υπάρχουν εκπρόσωποι που θα φέρουν πολιτικές ευθύνες και θα μπορούν να διεξάγουν τις συζητήσεις αυτές. Και αυτός λοιπόν είναι ένα σημαντικός παράγοντας ώστε να μπορούμε να συζητούμε τα θέματα αυτά με συνεργασία αυτών που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη. Εν συνόψη λοιπόν έχουμε διατηρήσει και εν μέρη μάλιστα επεκτείνει τις αρμοδιότητες επί του προϋπολογισμού. Έχουμε βελτιώσει σημαντικά τις πολιτικές δυνατότητες του Κοινοβουλίου. Έχουμε εξασφαλίσει την κοινοτική μέθοδο, διότι οι αρμοδιότητες παραμένουν εκεί όπου τις, όπου τις προβλέπει η συνθήκη. Δεν αποφασίζονται πλέον αυτά διακυβερνητικά, παραμένουν οι επίτροποι αρμόδιοι και ελπίζω ότι στην βάση αυτή θα δημιουργήσουμε μια ισχυρή εξωτερική υπηρεσία φτιάχνοντας έτσι μια πολιτική την οποία όλοι χρειαζόμαστε βεβαίως ο καθένας από εμά και όλοι μαζί θα την είχαμε φτιάξει διαφορετικά και πολύ καλύτερα αλλά μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για συνεργασία 3,5 θεσμικών οργάνων, αφού η κυρία Άστον είναι μισό θεσμικό όργανο για την ώρα ακόμα. Πρόκειται για ένα συμβασμό που ήταν σημαντικό να επιτευχθεί. Εγώ κατανοώ τι και του συναντέλφου που θα έρθουν και θα πούν δεν είναι σωστό το ένα ή δεν είναι σωστό το άλλο ή εδώ υπάρχει μια σάφια κτλ. Μέχρι ότου να θέσουν σε κίνδυνο ολόκληρο το οικοδόμημα αυτό. Και βέβαια θα υπάρχουν ελλείψεις και βέβαια θα υπάρξουν ανάγκες διευκρινήσεων. Αλλά όπως είπα πρόκειται για συμβασμό. Και το όλα ή τίποτα δεν υπάρχει όταν διαπραγματεύονται μεταξύ τους τέσσερα θεσμικά όργανα. Αυτό που χρειάζεται είναι να εξασφαλιστεί μια σωστή ισορροπία. Η κατάσταση τώρα για το Κοινοβούλιο είναι καλύτερη από ότι αν δεν είχαμε την συμφωνία αυτή. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερη ακόμα. Το δέχομαι. Αλλά είναι πάντως καλύτερη από αυτή που ισχύει τώρα. Και αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Και ακούγοντας πίσω μου τον αγαπημένο μου υποβολέα Σάριους Βόλσκι, τα τελευταία, τους, τε, τελευταίες, μην, τους τελευταίους μήνες τάχθηκε υπέρ μια ισότητα των φίλων Διορθώνω, διορθώνω. Γεωγραφική ισότητα. Πάλι τα μπερδεύω αυτά τα δύο. και αυτό το δέχτηκε στις 3 Μαΐου το Συμβούλιο μετά από δική μας πρόταση και έχει επεκταθεί μπαίνει και στις αιτιολογικές σκέψεις ότι οι χώρες μέλη που μειονεκτούν πρέπει να προτιμηθούν και αν μέχρι το 2013 δεν έχει επιτευχθεί η ισότητα αυτή θα πρέπει στην review phase να επανεξεταστεί δεν είναι το κείμενο αυτό τόσο λαμπρό όσο αυτό που είχε γράψει ο Γιάτσεκ Σάριου Βόλσκι, αλλά κατά το περιεχόμενο, κατά το ουσιώδε περιεχόμενο, είναι αυτό περίπου που χρειαζόμασταν. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να είμαστε σχετικά τουλάχιστον ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ. Λυπούμε μόνο που δεν είμαι νεότερος και δεν μπορώ να κάνω αίτηση να υπηρετήσω στη νέα αυτή υπηρεσία. μία διευκρίνηση σε αυτό που είπε ο κύριος Μπροκ. Μία νέα καριέρα στην υπηρεσία είναι ανοιχτή για όλους, φτάνει να παραμείνει το ευρώ. Θα ζητήσω τώρα από τον κύριο Γκουαλτιέρη που συμμετείχε στις θεσινές συζητήσεις να λάβει το λόγο και μετά θα δώσω το λόγο στους συζητητές. Σαλαφράνκα, Νέιτς, Τάνοκ και μετά Βόλσκι, Γιανιέζ, Λουέζινγκ και η κυρία Λούνατσεκ είναι η συγγήτρια επίσης. Μπορώ να μιλήσω ως ηγητής γιατί πρέπει να πάω στην κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία για το κοσυφοπαίδιο. Ναι, ναι. Ο κύριος Γκουαλτιέρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ξεκινώ από τις τελευταίες σκέψεις του συναδέλφου Μπροκ. Πρόκειται για έναν συμβιβασμό μετά από μία διαπραγμάτευση διαφόρων θεσμικών φορέων, σε μία διαπραγμάτευση με βάση μία διαδικασία διαβούλευσης. Αυτό προβλεπόταν για το Κοινοβούλιο και αυτό θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη στην αποτίμηση του αποτελέσματος. Αρκεί να συγκρίνουμε τις δύο στήλες του γράφου, δηλαδή την αρχική πρόταση άστον και το, την έκβαση της τελικής διαπραγμάτευσης για να δούμε ότι η διαβούλευση αυτή Η δυνατότητα διαβούλευσης, διαβούλευσης χρησιμοποιήθηκε σωστά από το Κοινοβούλιο στα πλαίσια μιας διαδικασίας συναπόφασης για κάτι το οποίο δεν ήταν μετατρέψιμο εξ αρχής. Νομίζω λοιπόν ότι ως προς τη μεθοδολογία, την όλη διαδικασία, δηλαδή φτάσαμε σε ένα πολύ καλό και εύλογο αποτέλεσμα. Ως προς την ουσία, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία. Αποφύγαμε έναν διτό κίνδυνο το να έχουμε μία μικρή υπηρεσία και καθόλου φιλόδοξη, έτσι ώστε να υπάρχει ένα εγκάρσιος διαχωρισμός μεταξύ διαφόρων μηχανισμών γεωγραφικής υφής. Άρα θα είχαμε μία υπηρεσία που δεν θα μπορούσε να συνδράμει στην συνοχή της εξωτερικής πολιτικής ή να έχουμε μια υπηρεσία που να είναι μακριά από την κοινοτική μέθοδο. Εμείς καταβάλαμε προσπάθεια για να έχουμε μια φιλόδοξη υπηρεσία με ευρείες αρμοδιότητες και παράλληλα συνδέοντας ε, αυτή, αυτό το φορέα με την κοινοτική μέθοδο. Άρα χρησιμοποίησαμε το άρθρο για τον προγραμματισμό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής και ως προς τη διαχείριση κρίσεων βλέπουμε ότι στην δήλωση για τη διάρθρωση της υπηρεσίας βλέπουμε ότι η πτυχή αυτή λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, δηλαδή διαχείριση κρίσεων και οικοδόμηση ειρήνης, peace building. έτσι ώστε να δούμε και τον διακυβερνητικό χαρακτήρα και το στρατιωτικό με το μη στρατιωτικό σκέλος. Καταφέραμε λοιπόν να περιορίσουμε τα προβλήματα καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που ενέταξαν την υπηρεσία αυτή εκτός Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα ως προς τον προϋπολογισμό διοικητικών εξόδων και λειτουργικών εξόδων. και για τη διαδικασία απαλλαγής και για τον ε, έλεγχο από το ελεγκτικό συνέδριο, την Όλαφ και ούτω καθεξής. Δηλαδή εντάξαμε όλους αυτούς τους μηχανισμούς και υπάρχει και η διάσταση του προσωπικού όπου είχαμε μία ενίσχυση για την γεωγραφική εξισορρόπηση του προσωπικού του διορισμού του προσωπικού που απομακρύνθηκε λίγο από την αρχική πρόταση, αλλά μπορέσαμε να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα, δηλαδή το μέγιστο δυνατό όσον αφορά τις δικές μας αρμοδιότητες. Δεν νομίζω ότι τα κράτη-μέλη έκαναν ό,τι μπορούσαν από πλευράς Συμβουλίου. και υπάρχει και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Υπάρχει η δήλωση των δέκα σημείων. Ιδιαίτερα το πρώτο και το δέκατο είναι άκρος σημαντικά. Και το δέκατο οδηγεί σε έναν επαναπροσδιορισμό της ΚΕΠΑ μέσα στα πλαίσια των προϋπολογισμών για τις διάφορες αποστολές για να έχουμε μία διαφάνεια ως προς το δημοσιονομικό έλεγχο. Τέλος, ως προς θέματα καθαρά χρόνου. Το θέμα της διαβούλευσης και των συμφωνιών θα πρέπει να αποτιμηθεί από τις πολιτικές ομάδες και μετά θα αποφασίσουμε κατά πόσο θα υποστηρίξουμε το όλο οικοδόμημα έτσι ώστε να εγκριθεί και από την Ολομέλεια του Ιουλίου. Η έκθεση δηλαδή Μπροκ Φερχόφστατ. Επίσης, θα πρέπει και η δική μας Επιτροπή να ενταχθεί σε αυτή τη διαδικασία προβολής του όλου θέματος έτσι ώστε να εγκριθεί τον Ιούλιο. Στο μέτρο του δυνατού. Τη στιγμή που οι πολιτικές ομάδες και οι επιτροπές θα αποτιμήσουν και θα αξιολογήσουν πλήρως τις εργασίες αυτές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο σχόλια θα ήθελα να κάνω σε σχέση με την ουσία και το όλο θέμα και ως προς τη διαδικασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου για την εργασία τους, η οποία οδήγησε σε σημαντικές προόδους και το πλέον σημαντικό είναι οι πολιτικές αρμοδιότητες της ύπατης εκπροσώπου. Διασφαλίσαμε αυτό το πλαίσιο αρμοδιοτήτων και διασφάλισής τους. Εδώ αποτείνομαι στους δύο διακεκριμένους συζητητές για να ρωτήσω κατά πόσο αυτός ο τετραμερής διάλογος οδήγησε σε ένα έγγραφο το οποίο μπορεί κάπως να αλλάξει μέσω τροπολογιών, γιατί αν δεν γίνεται αυτό, τότε χάνουμε χρόνο. Νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να γνωρίζουμε ότι πρόκειται για δύο ξεχωριστά εγχειρήματα. Η θέσπιση μιας πολιτικής συμφωνίας και το νομοθετικό έργο συναπόφασης που αφορά καθαρά το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της πολιτικής συμφωνίας, διότι οι αναθεωρήσεις του κανονισμού για το προσωπικό και του δημοσιονομικού κανονισμού θα λάβουν υπόψη τους όρους αυτής της συμφωνίας. Άρα, το μόνο που θα ήθελα να τονίσω είναι τη σημασία αυτής, αυτής της πολιτικής πτυχής της συμφωνίας. Εάν, όπως είπε ο κύριος Μπροκ, μπορούν να επέλθουν αλλαγές, θα ήθελα μετά από μία ταχεία ανάγνωση της ε, δήλωσης της ΥΠΑ της εκπροσώπου θα ήθελα να υποβάλω ορισμένα σχόλια τα οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή την πολιτική συμφωνία η οποία διεμήφθη με άλλα θεσμικά όργανα. Στο σημείο 1 μιλάμε για την ΚΕΠΑ και την πρόθεσή της και γίνεται λόγος για το, για το Προεδρείο. Νομίζω ότι μιλάτε για το διευρυμένο, για διευρυμένο Προεδρείο εδώ. Θα πρέπει να διευκρινιστεί. Στο 4 μιλάμε για μια ειδική ομάδα που θα έχει πρόσβαση στα έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα του Συμβουλίου. Λέμε ότι υπάρχει αυτή η διάρθρωση και η ρύθμιση, αλλά είπα ότι εκπρόσωπος θα προτείνει προσαρμογές σε σχέση με τις υπάρχουσες ε, διατάξεις. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτές τις τροποποίησεις και δεν αναφέρεται αυτό. Αυτή είναι μία δέσμευση που θα πρέπει να αναλυφθεί από την ύπατη εκπρόσωπο, διότι αυτό δεν είναι μονόδρομος. Στο 5 μιλάμε για την παρουσία των επικεφαλής αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα ως προσχέσεις με χώρες όπου έχουμε ε, σημαντικές ε, σχέσεις. Δεν θα πρέπει να μιλάμε για άτυπες informal εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να διαγράψουμε αυτή τη λέξη που δεν προδικάζει την έκβαση του όλου εγχειρήματος, αλλά ε, αν η όλη διαδικασία δεν είναι ικανοποιητική, δεν θα πρέπει τότε να έχουμε μόνο άτυπες ε, συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Το τελευταίο άρθρο δεν είναι σαφής οι φιλοδοξίες του Κοινοβουλίου, διότι στην Ολομέλεια μιλήσαμε για την, υπηρεσία, για την ύπαρξη μιας υπηρεσίας όπου θα πρέπει να υπερισχύει η κοινοτική μέθοδος. Και έγινε λόγος για το εν τρίτον το οποίο θα αποτελείται από διπλωμάτες, εν τρίτον από το Συμβούλιο και εν τρίτον από την Κομισιόν. Δηλαδή το 60% θα είναι υπάλληλοι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Δηλαδή το Συμβούλιο έχει 200 περίπου ε, υπαλλήλους, ενώ η Επιτροπή έχει τουλάχιστον 20.000. Ε, θα πρέπει λοιπόν όταν μιλάμε για το 1 τρίτον να συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Δηλαδή ε, μιλάμε για ένα 60% και ένα 30%. Υπάρχει ένα 10% που παραμένει στον αέρα. Θα ήθελα να ξέρω τι σκοπό έχουν οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου. Ως προς την διαδικασία είδαμε ότι η ύπατη εκπρόσωπος έκανε μία δήλωση ενώπιον της Ολομέλειας. Θα ήθελα αυτή η δήλωση να αλλάξει όπως πρότεινα και επειδή θα πρέπει να εγκριθεί αυτό το πλαίσιο τον Ιούλιο από εμάς, θα θέλαμε μία πρόταση ψηφίσματος έτσι ώστε να δούμε και το νομοθετικό περιεχόμενο της πρότασης. Θα ήθελα μία διασάφηση ως προς τις προθεσμίες. Ο κύριος Μπρόκ μας είπε ότι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων θα υποβάλει τροπολογίες μέχρι τη Δευτέρα και μας είπε ότι η Επιτροπή θα μας παρουσιάσει την πρότασή της για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αύριο. Θα γίνει παρουσίαση από τον κύριο Φερχόφστατ. Θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε και την τελική έκβαση, δηλαδή μπορούμε να συζητήσουμε μετά την τελική έκβαση των συζητήσεων. Η κυρία Νέιτς. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, καταρχάς να συγχαρώ τους διαπραγματευτές για τα αποτελέσματα που πέτυχαν. Θεωρώ ότι η επιτυχία ήταν μεγαλύτερη από αυτή που θα μπορούσαμε να περιμένουμε λίγο πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων, όταν ε, υπήρχαν πολύ περισσότερες διαφωνίες. Σας υπενθυμίζω ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για όλα τα θέματα που είχαν να κάνουν με τον προϋπολογισμό και τον έλεγχο του Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό. Συγχαρητήρια λοιπόν στους τρεις διαπραγματευτές. Ήδη αναφέρθηκαν κάποια θετικά σημεία, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι 60% του προσωπικού της υπηρεσίας θα προέρχεται από τις εθνικές δημόσιες υπηρεσίες. Η διασφάλιση ότι οι επικεφαλής αντιπροσωπιών θα μπορούν να εμφανίζονται ενώπιόν μας πριν αναλάβουν τα καθήκοντα που θα προβλέπει η εντολή τους, κάτι που θα μας επιτρέπει έλεγχο των αποστολών. Επίσης, η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον διορισμό των επικεφαλής των αποστολών. Αυτά είναι όλα θετικά σημεία. Επίσης, θετικό σημείο είναι το γεγονός ότι η διαχείριση κρίσεων και η οικοδόμηση της δημοκρατίας αναφέρονται στην απόφαση. Βλέπουμε επίσης ότι στο πλαίσιο της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης θα υπάρχει και ένα τμήμα που θα βοηθάει την ύπατη εκπρόσωπο στη σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως βλέπουν οι συνθήκες όσον αφορά την πολιτική ευθύνη του Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θεωρώ ότι αυτός θα είναι ένας τρόπος να διασφαλίσουμε ότι οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες θα μπορούν να βοηθούν και τις εθνικές αντιπροσωπείες, κάτι που ήδη γίνεται. Η πολιτική μας ομάδα θεωρεί λοιπόν ότι τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα από ό,τι αναμέναμε στην έναρξη της διαδικασίας. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, συμφωνούμε ότι στο μέτρο του δυνατού αυτή η σημαντική απόφαση πρέπει να ληφθεί ήδη στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Βεβαίως όλα θα εξαρτηθούν από την ταχύτητα με την οποία θα λάβουμε το κείμενο και το κατά πόσο θα μπορέσουν να το εξετάσουν γρήγορα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές. Διαφορετικά θα μπορούσαμε να επιλέξουμε τη λύση Σαλαφράνκα που επίσης ακούγεται καλή, δηλαδή η έγκριση ενός ψηφίσματος όπου θα συμπεριλαμβάνουμε όλα τα σημαντικά στοιχεία. Το ιδανικό βεβαίως θα μπορούσαν να θα έπρεπε να ήταν έγκριση τον Ιούλιο στην Ολομέλεια. Θα χρειαστεί πολύ καλή θέληση, αλλά νομίζω ότι υπάρχει. Τέλος, να πω ότι ίσως είναι αναπόφευκτο, αγαπητοί συνάδελφοι, η υλοποίηση αυτών των νέων θεσμικών οργάνων που προβλέπονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας και τα νομοθετικά κείμενα τα σχετικά, τα σχετικά εδώ με την ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης, θα μπορέσουν να αποτελέσουν ε, και έναν τρόπο να καλύψουμε το κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη διεθνή παρουσία της Ένωσης. Και ελπίζω το κενό να καλυφθεί το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Να σας ενημερώσω ότι το σημείο που ακολουθούσε αυτή τη συζήτηση, παρουσίαση του κυρίου Κούπερ δηλαδή, αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση και ευχαριστώ τον κύριο Κούπερ για την κατανόησή του και του ζητώ συγγνώμη γιατί θέλουμε χρόνο στη διάθεσή μας για τη συζήτηση αυτού του σημαντικού θέματος. Κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ ονόματος των Πρασίνων θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους τρεις διαπραγματευτές, οι δύο είναι παρόντες, για την εργασία τους εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, ήταν δύσκολες οι συζητήσεις και όπως και άλλοι έτσι και εγώ στην αρχή δεν περιμέναμε να καταφέρουμε τόσα πολλά. Το ελπίζαμε βεβαίως, προσβλέπαμε σε αυτό, αλλά υπάρχουν ε, πολλά στοιχεία που δεν ήταν προγραμματισμένα, δεν προβλέπονταν και η ομάδα μας θεωρεί ότι σε πολλά θέματα υπάρχει πρόοδος, διαφάνεια, πρόσβαση σε πληροφορίες. Οι δύο δηλώσεις ε, όπου η Άστον είπε ότι θα δημοσιευθούν στην επίσημη εφημερίδα οι δηλώσει ενώπιον τη ολομέλεια που τους προσδίδει πολύ πιο επίσημο χαρακτήρα από μία απλή δήλωση. Και επίσης τρία πράγματα ήταν πολύ σημαντικά για μας. Το πρώτο ήταν τα χρηματοδοτικά, χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία είναι υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για αυτούς που εργάζονται σε αναπτυξιακούς οργανισμούς. Δηλαδή, η ανάπτυξη δεν πάει κάτω από τις ε, εξωτερικές υποθέσεις. Δεν αντιτάσσονται τα δύο. Στην αρχική πρόταση Άστον και στην πρόταση του Συμβουλίου δεν υπήρχε τίποτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και καταφέραμε να έχουμε ένα τμήμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην έδρα αλλά και σε κάθε αντιπροσωπεία να υπάρχει ένα γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όποιος έχει ε, εργαστεί για την κοινωνία των πολιτών πριν γίνει πολιτικός, γνωρίζει ότι αυτές οι οργανώσεις, οι περασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κοινωνία των πολιτών, εκείνοι που είναι υπέρ της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας, ε, θέλουν να ξέρουν ότι υπάρχουν ένα ή δύο πρόσωπα στα οποία μπορούν να αποτανθούν, θα εισακουστούν και θα τους βοηθήσουν έτσι ώστε να εφαρμοστούν τα δικαιώματά τους για το προσωπικό, την επάνδρωση, ε, έχει σημασία η ισότητα, η εκπροσώπηση των δύο φύλων, γιατί στις εξωτερικές υποθέσεις και στη διπλωματία ε, δυστυχώς δεν υπάρχει ισότητα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει επί του παρόντος και πρέπει να εξασφαλιστεί. Α, στον Καναδά, εντάξει, ίσως στον Καναδά, ναι. Το ξέρω αλλά μία χώρα δεν αρκεί. Θα πρέπει να μιλάμε για εν τρίτον καταρχήν, αλλά καλύτερα 50-50. Να εξασφαλίσουμε την ε, ισότητα πρόσβασης των δύο φύλων και τη γεωγραφική κατανομή, που να είναι δίκαιη για να εκπροσωπηθούν όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης, επιτελέστηκε κάποια πρόοδος ως προς την ε, νέα κατάλληλη διάρθρωση για τις αποστολές ε, ΚΕΠΑ στην Επιτροπή. Δηλαδή, η ΚΕΠΑ δεν θα αφορά μόνο το Συμβούλιο, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς ως πράσινοι θα θέλαμε η διαχείριση των ε, κρίσεων να έχει δεσπόζοντα χαρακτήρα, αλλά η Κάθριν Άστον υποστηρίζεται αρκετά έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πρωταρχικό ρόλο στην διαχείριση των κρίσεων και την οικοδόμηση της ειρνευτικής διαδικασίας. Αυτά είναι τα θετικά στοιχεία. Θα θέλαμε να είχαμε και μόνιμη παρουσία πολιτικών, αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν. Δεν θα υπάρχει μία ε, πολιτική Γενική Γραμματεία. Ε, πετύχαμε αρκετά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ως προς το χρονοδιάγραμμα, νομίζω ότι για να προχωρήσουν τα πράγματα θα έπρεπε να επέλθει συμφωνία κατά την Ολομέλεια του Ιουλίου. Εμείς θα το υποστηρίξουμε ως προς τον προϋπολογισμό και το καθεστώς του προσωπικού θα πρέπει να ακολουθήσουμε την κοινοβουλευτική διαδικασία έτσι ώστε να το επιτύχουμε μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις με την Άστον και επ' αυτού. Δεν είναι επίκαιρο, αλλά είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Ευχαριστούμε. Επειδή και εμείς είμαστε άνθρωποι ε, ως βουλευτές θα πρέπει να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα παντού και σε όλους τους τομείς ε, Τάνοκ. Έχουμε μία κάπως διαφορετική άποψη στην ομάδα μου, αλλά θα ήθελα να συγχαρώ τους κυρίους ε, Μπροκ, Φερχόφστατ και Γκουαλτιέρη για την εξαιρετική τους εργασία, ενισχύοντας το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί αυτό που αρχικά ήταν η αρχική όθηση είχε δοθεί από το Συμβούλιο. Ορισμένες ε, ιδέες υλοποιήθηκαν. Η Βαρόνη Άστον θέλει να αφήσει ένα κληροδότημα και βεβαίως αυτή είναι η βαριά εργασία η οποία θα πρέπει να επιτελεστεί μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ίσως είμαι υπερβολικά αισιόδοξο, αλλά με εκπλήσει αυτή η ιονή συμφωνία διορισμών, διαδικασίας διορισμών. Αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να διορίσει ειδικού εκπροσώπου ή διπλωμάτες. Δηλαδή δεν πρόκειται για εξουσίες καθαρά κοινοβουλευτικέ για μας. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να αρκεστούμε στη συναπόφαση, στι διαδικασίε συναπόφασης ε, δυνάμει της ε, συνθήκης της Λισαβόνα και για την ΚΕΠΑ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η εξέλιξη σε ένα σημείο του εγγράφου μιλάτε για δημοσιονομικό έλεγχο για τις δραστηριότητες ΚΕΠΑ. Μιλάτε για το μη στρατιωτικό σκέλος, γιατί το στρατιωτικό καλύπτεται από τα κράτη-μέλη. Δεν γίνεται λόγος για τους εθνικούς βουλευτές σε σχέση με τον έλεγχο της ΚΕΠΑ που είναι ύψης της σημασίας ιδιαίτερα μετά την διάλυση της ε, Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί διαφορετικά θα απομακρυνθούν τα εθνικά κοινοβούλια στον έλεγχο της ε, κοινή ε, δράσης εξωτερικής πολιτικής. Ως προς την άρση των μόνιμων εκπροσώπων των μόνιμων υπουργικών θέσεων, αυτό με εκπλήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει το ότι επανέρχονται υπουργοί εξωτερικών είναι κάτι πολύ καλό. Αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπε η κυρία Λούνατσεκ, θα υπάρχουν γεωγραφικά, γεωγραφική, θα υπάρχει γεωγραφική κατανομή γραφείων. Ως προς τη γεωγραφική εξισορρόπηση που απασχολεί τον κύριο Σάριους Βόλσκι και πολλούς άλλους, εγώ νομίζω ότι η αξιοκρατία έχει μεγαλύτερη σημασία και όχι η γεωγραφική εξισορρόπηση. Γιατί το κριτήριο είναι η αξιοκρατία, όχι η γεωγραφική κατανομή. Μιλάμε δηλαδή για γεωγραφική εξισορρόπηση, αλλά ζητάμε για το ότι η σύνθεση θα πρέπει να μείνει παρά, να, μην, να μην ε, αλλάξει καθόλου, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν υπάρχει κανένα μέλος από πλευράς Γαλλίας ή Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτούς τους ε, διορισμούς και δεν γίνεται λόγους για, τις, ε, για τα προξενία ως προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θα θέλαμε να ξέρουμε τι θα γίνει σε σχέση με τα εθνικά προξενία ως προς τα προξενία που θα εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ο κύριος Βιγγένιν, ο συντονιστής, ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Βλέπετε ότι υπάρχει ευρία συνένεση στην αίθουσα για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Στηρίζουμε πλήρως την θέση του κυρίου Γκουαλτιέρη και θεωρούμε πολύ σημαντικό το να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τον Ιούλιο. Καταλαβαίνω ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο. Όμως το έχουμε ήδη συζητήσει. Είχαμε πει αν καταλήξουμε σε συμφωνία θα πρέπει να το προσπαθήσουμε. Και παρόλο που κάποια θέματα ίσως ε, θα χρειάζονταν περισσότερη συζήτηση, για παράδειγμα ο κανονισμός προσωπικού, Θεωρούμε ότι πρέπει να λήξει το θέμα μέχρι τον Ιούλιο για να μπορέσει να λειτουργήσει η υπηρεσία το φθινόπωρο. Ευχαριστώ κύριο Βόλσκι. Ζητώ συγγνώμη από τον Έλμαρ Μπροκ που θα ξανακούσει αυτά που του έχω ήδη πει. Πρώτα, επαναλαμβάνω πρώτα ότι πρέπει να επενέσουμε και να συγχαρούμε τους εκπροσώπους μας οι οποίοι πέρασαν μέσα από αυτή τη διαδικασία δύσκολων συνομιλιών με την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω και αν είναι πράγματι 3,5 τα θεσμικά όργανα, γιατί εγώ θεωρώ το κοινοβούλιο 1,5 θεσμικό όργανο, άρα μας κάνει τέσσερα. Και ειδικά με σένα, Έλμαρ, επικεφαλής, σίγουρα είμαστε, ε, γίνονται τέσσερα τα όργανα. Τώρα, πόσο προχωρήσαμε στην κοινοτικοποίηση, όπου εγώ πραγματικά καταχάρηκα από αυτή την επιτυχία μας. Συνολικά υπάρχει πρόοδος όσον αφορά και ε, την, ε, από, την κατανομή ε, ευθυνών, την accountability. Εάν πρόκειται πάντως να κρίνουμε για το που βρισκόμασταν πριν από τη Μαδρίτη και που βρισκόμαστε τώρα μετά την Μαδρίτη, θα ήταν καλύτερα να κάνουμε ένα πίνακα των διαφόρων εγγράφων. Και θα παρακαλέσω τη Γραμματεία να συγκρίνει ε, το έγγραφο της 3ης Μαΐου με αυτό που προέκυψε μετά τη Μαδρίτη. Τώρα το ποτήρι μου φαίνεται μισογεμάτο, το μπουκάλι, αλλά δεν είναι εντελώς γεμάτο, ναι. Έξι χρόνια κι εγώ ε, στην ΑΦΕΤ είδα ότι η Επιτροπή μας ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξη. Πάντοτε θαύμαζα τον Έλμαρ Μπροκ διότι αγωνιζόταν και πάντοτε και πάνω από τα κιλά του σε κατηγορίες δηλαδή μεγαλύτερων βάρων από τα κιλά του ας το πω έτσι και από τα δικά μου αγωνιζόταν πάντοτε δεν θα πω τώρα με ποιον πάντως για μεγαλύτερο ρόλο της Επιτροπής ΑΦΕΤ αλλά και του Κοινοβουλίου στις εξωτερικές υποθέσεις και εξακολουθούμε και έχουμε βάρος στις ε, διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ας εκμεταλλευτούμε τη βαρύτητα αυτή που έχουμε ώστε να γεμίσουμε το μπουκάλι ακόμη περισσότερο. Όντας τόσο θετικός και συγχαίροντας ε, τους ε, Μπροκ και Βεχόφστατ, πρέπει ωστόσο να σημειώσω και δύο ελλείψεις. Δεν έχουμε πολιτικούς μέσα εκεί και ούτε οι ε, διαδοχικές προεδρίες θα είναι οι κατάλληλοι συνομιλητές ε, αυτοί που έρχονται κάθε έξι μήνες και μας λένε κάνουν ό,τι μπορούν. Καλύτερα θα ήταν να έχουμε ε, μόνιμους πολιτικούς ε, αναπληρωτές της Άστον και όχι αλληλοδιαδεχόμενους ανά εξάμεινο. Τώρα, η εξωτερική υπηρεσία θα πρέπει να είναι από την αρχή με εξωτερική υπηρεσία των 27 και όχι των 15, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος αυτός. Οι βελτιώσεις είναι σημαντικές και για την ε, συμμετοχή όλων των χώρων μελών. Αλλά αυτό το λέει ήδη το άρθρο 27 του καταστατικού των υπαλλήλων της Κομισιόν. Καλά είναι που τα λέει λοιπόν εδώ για την ισότιμη εκπροσώπηση όλων των χωρών, αλλά δεν είναι και τίποτα το νέο. Τώρα, η, φάση αναθεώρηση του 2013. Είναι καλό που λέει ότι θα επανεξεταστεί το 2013. Τώρα, γιατί να ικανοποιούνται οι στόχοι κατά το 25% μόνο των νέων χωρών μελών. Το ίδιο θα ισχύει και σε τρία χρόνια. Εάν μετά από πέντε χρόνια ισχύω του κανονισμού έχουμε φτάσει στα 25% μονάχα στην ΡΕΛΕΞ, χωρίς αυτό τον κανονισμό θα είχε υπάρξει ε, πρόοδος και σε πόσα χρόνια. Καλύτερα λοιπόν, αλλά όχι αρκετά. Από τα απομνημονέματα του Σαμονέ λέω ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς τον άνθρωπο ή χωρίς ανθρώπους σαν τον Μπροκ, ας το πω έτσι. Ομ, ανθρώπους, αλλά και άνδρες, άνδρες ή γυναίκες. Σε πάση περιπτώσει, Ζαμονέ τα είπα αυτά τα πράγματα. Δεν μου ζητάτε να αλλάξω τώρα τα πνευματικά του Ζαμονέ. Άρα και τίποτα δεν έχει διάρκεια χωρίς θεσμούς. Αν το μεταφράσω στα αγγλικά θα έλεγα, πάλι ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς ανθρώπους, γυναίκες ή άνδρες, αλλά και τίποτα δεν έχει διάρκεια ή δεν είναι βιώσιμο χωρίς θεσμούς. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε τότε τον 241 κάθετος 2 του 2004, τον κανονισμό αυτό δηλαδή, που προβλέπει 36 επικεφαλής αντιπροσωπιών από 5 πολιτικές ομάδες από 15 χώρες μέλη, όχι μόνο τις νέες, αλλά και τη Γερμανία και την Ιταλία, που εκπροσωπούν 261 βουλευτές. Όλοι αυτοί, οι όλοι μας, ας ψηφίσουν τους συμβασμούς που επιτεύχθηκαν και ας τους εγκρίνουν. Δεν είναι το τέλος εδώ, είναι μόνο η αρχή, θα συνεχιστεί η διαδικασία και εγώ ως συντάκτης της γνωμοδότησης της ΑΦΕΤ για το καταστατικό του προσωπικού αναμένω τη συνεργασία του Συμβουλίου. Ναι, α το πω έτσι. Εν τέλει, ποιο θα είναι το νομικό καθεστώ, ή μάλλον ποιο είναι το νομικό καθεστώ και η δεσμευτικότητα της συμφωνίας αυτή, Είναι και δεσμευτική και για τον διάδοχο της Λέιδη Άστον. Και θα μπουν και όλα στο κείμενο αυτό και της IIA και οι δύο κανονισμοί επίσης. Και από εδώ στον κύριο Τάνοκ. Άλλο τα προσόντα, άλλη η, γεωγραφική ισορροπία. Σας ευχαριστώ. Θα μείνουν οι μεταφραστές μέχρι τις 7 παρατέταρτο. Έχουμε ακόμα ορισμένους που ζητάνε το λόγο. Μετά θα ζητήσω τον κύριο Μπρόκ να συνοψίσει τη συζήτηση. Ο κύριος Ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα να μπω στην ουσία της συζήτησης. Έχει υπάρξει συνένεση και συμφωνώ με τους ε, παρεμβαίνοντες και τις παρεμβαίνουσες. Θα ήθελα να συγχαρώ τους ε, διαπραγματευτές. Εγώ είμαι σοσιαλδημοκράτης και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γουαλτιέρη, τον Ρομπέρτο Γουαλτιέρη που μας εκπροσώπησε πολύ καλά, αλλά και τους Μπροκ και Φερχόφστατ. Νομίζω ότι προχωρήσαμε αρκετά ε, σε σχέση με τον ευρωσκεπτικισμό που υπήρχε λίγες μήνες πριν. Φτάσαμε σε έναν εξευρωπαϊσμό της υπηρεσίας αυτής και βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ασχοληθεί με το δημοσιονομικό κανονισμό για τον έλεγχο αυτής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ζήτησα το λόγο ως εκπρόσωπος ε, της διάσκεψης των Προέδρων από τις αντιπροσωπείες και επίσημα θα ήθελα να πω προς τους ε, κυρίους Μπροκ και Γκουαλτιέρη ότι στις 7 ε, Ιουλίου θα πρέπει να εξηγήσουν σε όλους τους εκπροσώπους το πώς λειτουργεί αυτή η υπηρεσία, το πώς θα λειτουργήσει αυτή η υπηρεσία. και πώς μπορούν να βρουν μια καλή συμμαχία για να λειτουργήσει έμπρακτα αυτή η υπηρεσία. Δηλαδή στη ε, διάσκεψη, Προέδρων των Διεθνών Αντιπροσωπιών σε 7 Ιουλίου θα πρέπει να λογοδοτήσετε κατά κάποιο τρόπο. Η κυρία Λέζινγκ. Παρόλες τις βελτιώσεις που επιτεύθηκαν χάρη στην στεναρή στάση των βουλευτών μας και που σίγουρα χωρίς αυτήν δεν θα είχαν επιτευθεί, παρόλα αυτά στο όνομα της ομάδας της Ενωτικής Αριστεράς δεν μπορώ να συμμετάσχω σε αυτήν την χαρούμενη ατμόσφαιρα που διαδίδεται εδώ. Για μας με την συμφωνία αυτή της Μαδρίτης μειώνονται οι ελπίδες σαφώς για μια ειρηνική εξέλιξη των εξωτερικών σχέσεων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεν θέλουμε συνένωση στρατιωτικών και μη στρατιωτικών δομών. Για μας αυτά είναι απαράδεκτα. Ούτε υπάρχει καμία υπηρεσία εξωτερικής δράσης στον κόσμο που να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η πραγματική μη στρατιωτική εξωτερική δράση ως πραγματική επιλογή απομακρύνεται. Και μία πτυχή που δεν συζητείται εδώ πια είναι και η συμμετοχή έμεσα έστω των μυστικών υπηρεσιών στην υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Βέβαια θα αρκεστώ σε αυτά γιατί τα έχω ξαναπεί εδώ στο Κοινοβούλιο. Η κριτική μας παραμένει πάντως. Ερώτηση προς τον κύριο Μπρόκ είπατε ότι ο κύκλος εκείνων ο οποίος θα έχει πρόσβαση στο μέλλον σε εμπιστευτικά έγγραφα διευρύνεται. Η ερώτησή μου είναι εάν θα περιλάβει αυτό και βουλευτές της Ενωτικής Αριστεράς. Ευχαριστώ, κύριος Ξύπλης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρα. Θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους που συνεχάρηκαν τους διαπραγματευτές, ειδικά τον κύριο Μπρόκ. Θέλαμε πολλά να επιτύχουμε από την αρχή. Το είχαμε συζητήσει εκτεταμένα το θέμα στην ΑΦΕΤ και γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα που επιτύχαμε πολλές από αυτές τις επιθυμίες μας. Όπως είπα και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Χαίρομαι που βλέπω ότι θα υπάρχει παντού ένα άτομο υπεύθυνο για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με κυβερνητικές οργανώσεις κτλ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ειδικά για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα άτομα που διώκονται. Είναι μια εγγύηση ότι σε κάθε αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα υπάρχει ένα άτομο που θα μπορεί να τους μιλήσει, να είναι το σημείο επαφής τους. Βεβαίως από ό,τι φαίνεται δεν επιτύχαμε το 100% των στόχων μας υπάρχει ισότητα των φύλων, θέλαμε και γεωγραφική ισότητα, οπότε εδώ θα συμφωνήσω με τους άλλους συναδέλφους. Βεβαίως θα υπάρξει αναθεώρηση το 2013. Αλλά σας υπενθυμίζω ότι όταν εμείς ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχαν περιορισμοί στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Στην αρχή ελπίζαμε ότι με κάποια αναθεώρηση θα μειώνονταν αυτοί οι περιορισμοί νωρίτερα, αλλά εξαιτία των οικονομικών προβλημάτων δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη και για την γεωγραφική ίση εκπροσώπηση. Ένα άλλο θέμα, τη σαφήνεια των διατυπώσεων, ειδικά όσον αφορά τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων και το αριθμό του προσωπικού. Είναι απαραίτητο να υπάρξει αυτή η σαφήνεια γιατί όπως είπε και ο κύριος Αλαφράγκα διαφορετικά θα περιπλακούν πολύ τα πράγματα. Και μία ερώτηση προς τον εισηγητή. Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε μια πιο σαφή όσον αφορά την Τρόικα. τι ακριβώς θα ισχύει. Θα υπάρχει εντολή που θα δίνει η ύπατη εκπρόσωπος. Ή θα χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο είδος συντονισμός που θα μπορούσε να ικανοποιήσει και το Κοινοβούλιο και το Υπουργείο Εξωτερικών της εκάστοτε Προεδρίας. Ένα τελευταίο σχόλιο. Θεωρώ ότι τα εθνικά κοινοβούλια δυστυχώς εξαιρέθηκαν από την διαδικασία και πρόκειται να ακούσουμε πολλές επικρίσεις γι' αυτό γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται πουθενά στη διαδικασία. Εδώ συμφωνώ με τον ε, κύριο Τάνοκ που επίσης το ανέφερε. Θα σας μιλήσω και από την εμπειρία μου ως εθνικός βουλευτής. Θυμάμαι ότι είχαμε πολλές προσδοκίες που δεν επιβεβαιώνονταν πάντα. Ευχαριστώ κύριος Μπρόκ. Αν τα καταφέρατε σε 7 λεπτά... Θα προσπαθήσω πρόεδρε. την δήλωση των διαπραγματευτών λέγεται ότι κάθε πλευρά θα προσπαθήσει τώρα να επιτύχει την υποστήριξη εντός του θεσμικού της οργάνου. Αυτό είναι σαφές. Δεύτερο είναι σαφές επίσης ότι η νομοθετική διαδικασία επηρεάζεται περιορισμένα από την συμφωνία. Ειδικά διότι έχει διαγραφεί το άρθρο για το καταστατικό των υπαλλήλων της υπηρεσίας. Ε, βεβαίως υπάρχει δυνατότητα τροποποιήσεων. Όταν όμως έχει επιτευχθεί ένα πολιτικό πλαίσιο μιας συμφωνίας, είναι σωστό να προσπαθήσει κανείς να τηρήσει το πλαίσιο αυτό. Διότι εάν το τροποποιήσει δίνει το δικαίωμα στην άλλη πλευρά να προβεί και αυτή σε τροποποίηση της θέσης της. Ενώ εμείς ενδιαφερόμαστε να υπάρξει πλειοψηφία του σώματος. Για την πολιτική δήλωση αναφέρεται στα προεδρία της, ε, της Επιτροπής Εξωτερικών και της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Και μόνο από κοινού μπορούν να γίνουν οι αλλαγές. Και αυτά μόνο για περιπτώσεις που άπτονται των προϋπολογισμών. Για την κοινή εξωτερική πολιτική πολιτική ασφάλειας, όπου απριόρι θίγονται οι συγκεκριμένες αυτές επιτροπές. Πάντοτε εμείς είχαμε να συνεργαστούμε με την Επιτροπή Προπολογισμών. Και αυτό με ενοχλούσε, διότι καταρχήν για τα εξωτερικά, για τι εξωτερικέ σχέσει, αρμόδια είναι η Επιτροπή Εξωτερικών. Τώρα, για την εξέταση εμπιστευτικών εγγράφων και για αυτή την πενταμελή επιτροπή. Αυτό είναι διαθεσμική συμφωνία και η διαθεσμική συμφωνία αλλάζει μόνο αν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρέ τη διαθεσμική συμφωνία. Άρα πάλι αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρί την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια ε, διαθεσμική συμφωνία η οποία έχει συναυθεί εδώ και 5-6 χρόνια. Τώρα για τις ακροάσεις. Εμείς είχαμε δεχθεί όταν ήταν εδώ παρόν ο κύριος Αλμέιντα να, ότι, ότι υπήρξε ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων και κλεισμένο των θυρών μεταξύ Αλμπερτίνη και Άστον. Και δεν θέλαμε να φύγει η λέξη ανεπίσημος διότι δεν πρόκειται για ακρόαση όπως αυτές προβλέπονται στην συνθήκη. Αλλά αφαιρέθηκε ο όρος in camera και κλεισμένο των θυρών δηλαδή. Καταφέραμε τέλο πάντων να αφαιρεθεί ο ένας από τους δύο όρους. Επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτα, γιατί και στις ανεπίσημες ανταλλαγές απόψεων υποβάλλεται επιστολή του Προέδρου στην ύπατη εκπρόσωπο για αξιολόγηση. Και αυτό λοιπόν το έχουμε εξασφαλίσει για το μέλλον. Τώρα για τα 60% αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπαμε τουλάχιστον 60% και τουλάχιστον ένα τρίτο προσωρινών υπαλλήλων από τις χώρες μέλη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει ένα περιθώριο που μπορεί να περιλαμβάνει για παράδειγμα στρατιωτικούς και αστυνομικού, οι οποίοι αποστέλλονται εδώ με αποστολές από τις χώρες μέλη. Όπως είπα, είναι τα ελάχιστα όρια αυτά, 60% και 1 τρίτο. Και 30% συγγνώμη. Και είπαμε το υπόλοιπο μπορεί να είναι μόνο για ειδικέ περιπτώσεις. Δεν θέλουμε να πλημμυρίσει η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων με φθηνό εντό αγωγών προσωπικών των χωρών μελών το οποίο πληρώνουν λιγότερο οι χώρες μέλη. Ενημερώσαμε κύριε Σαλαφράγκα σήμερα το πρωί τους πρόεδρους των πολιτικών ομάδων, τους εισηγητές. Έχουμε ενημερώσει ήδη σήμερα το πρωί την Επιτροπή, την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Αναπτύξεως και σήμερα το μεσημέρι στη μία η ώρα ενημέρωσα και διεξοδικά μάλιστα όλα τα μέλη του Λαϊκού Κόμματος που συμμετέχουν στην Επιτροπή Εξωτερικών. Οι συνομιλίες λοιπόν συνεχίζονται. Νομίζω ότι αρμόζει αυτό στην σημασία του θέματος. Για την κυρία Νάιτς Ευχαριστώ για τις σημειώσεις σας. Δεν ξέρω αν η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί απλά με ένα ψήφισμα. Είναι σημαντικό βέβαια να υπάρξει ψήφισμα όπου να κάνουμε ορισμένες διακριβώσεις και να ορίσουμε πώς κατανοούμε τα κείμενα, να βάλουμε ορισμένους ορισμούς μέσα. Και αυτό ισχύει και ειδικότερα για τον τομέα του προϋπολογισμού. Αλλά Μπορούμε να ρωτήσουμε και τον κύριο Σαλαφράνκα. Αυτό θα μας βοηθήσει και για το μέλλον και ιδίω για την political accountability. Στις χώρες μέλη δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα γιατί μέσα από τους αιώνες έχουν αυξηθεί οι αρμοδιότητε των κοινοβουλίων απέναντι στι κυβερνήσει. Ενώ εμεί είμαστε υποχρεωμένοι για να αποκτήσουμε δικαιώματα να περάσουμε μέσα από διαπραγματεύσει. Και βέβαια αυτέ οι διαπραγματεύσει παραμένουν πολιτικού χαρακτήρα, που αποτελούν πολιτικέ δεσμεύσει. Δεν είναι νομικά κείμενα για τέτοιε πολιτικέ δεσμεύσει, ούτε προβλέπονται μέσα στι συνθήκε. Πάντοτε θα έχουμε τη δυσκολία αυτή αλλά αυτή είναι και η μέθοδος την οποία πάντοτε εφαρμόσαμε μέχρι τώρα. Είτε με συμφωνία, είτε με αποδοχή δηλώσεως την οποία κάνει η άλλη πλευρά σε ένα συγκεκριμένο όργανο και περιλαμβάνεται μετά στα πρακτικά και το, το Συμβούλιο εγκρίνει μέσα στα πρακτικά του τις αποφάσεις των αποφάσεων, τις αποφάσεις μάλλον του Συμβουλίου και με τον τρόπο αυτό αποκτούν δεσμευτικότητα. Και να δούμε αν και εμείς έχουμε το ανάστημα να επιμείνουμε και να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα. Πώς θα ολοκλώσουμε τη διαδικασία κυρία Νάιτς, το είπαν και άλλοι, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Πάντως προτείνω να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις που χρειάζονται να καταθέσουμε σχέδιο ψηφίσματος. Προτείνω μάλιστα προληπτικά για την Τρίτη να βάλουμε προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, εάν θα τηρηθεί αυτή ή όχι αυτό, το βλέπουμε, αλλά προληπτικά ας το βάλουμε έτσι. Για την κυρία και ευχαριστώ και πάλι. Πράγματι, σωστά είπατε ότι δεν μπαίνουν στοιχεία τη πολιτική ανάπτυξη, τη πολιτική εξωτερικών κτλ. Γίνεται συντονισμό των πολιτικών αυτών όπω και πρέπει. Και νομίζω ότι είναι πολύ λογική αυτή η υπόθεση. Για τον κύριο Τάνοκ, πρώτη δωδεκάτου έναρξη της ε, δράσεω τη υπηρεσία. Εγώ θεωρώ ότι είναι δυνατόν αυτό, όντω. Δεν είναι μόνο θέμα του δημοσιονομικού κανονισμού, ούτε τόσο το θέμα του καταστατικού του προσωπικού, αλλά τι γίνεται με τον τροποποιημένο προπολογισμό του 2010. Περισσότερο από εκεί εξαρτάται. Ή κατά πόσον χρειάζεται να θεσπιστούν κάποιες μεταβατικές ρυθμίσεις που είναι βέβαια περίπλοκες. Αλλά δεν είναι δική μας υπόθεση αυτή εδώ. Εμείς αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργήσουμε τι προποθέσει για να μπορεί να λάβει απόφαση το Συμβούλιο. Και είπαμε μάλιστα και σήμερα, το συζητήσαμε και με του συζητητέ, ότι η απόφαση τη Ολομέλεια για τη staff regulation και τη financial regulation θα πρέπει να λαμβάνεται μετά από την απόφαση του Συμβουλίου. Ώστε εάν μας εξαπατήσει το Συμβούλιο να έχουμε δυνατότητα εμεί μετά να λάβουμε απόφαση. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση γιατί το τίμημα θα ήταν υψηλό για όλες τις πλευρές. Θα οδηγούσε άλλωστε σε περαιτέρω σημαντικές καθυστερήσεις. Εμείς θα επιμείνουμε στην δέσμη αυτή. Επιμείναμε και μέχρι τώρα και νομίζω αυτό μας βοήθησε στην διαδικασία. Ο έλεγχος του προϋπολογισμού τώρα αναφέρεται στο σύνολο του προϋπολογισμού της ΚΕΠΑ. Μέχρι τώρα είχαμε κάποια μειονεκτήματα, το γνωρίζουν οι αρμόδιοι του ελέγχου του προϋπολογισμού και διότι μέχρι τώρα αναμειγνύονταν το Συμβούλιο και η Προεδρία του Συμβουλίου και διότι υπήρχε συμφωνία κυρίων και μπορούσαν να τα ανακατέψει το Συμβουλίο. Τώρα όμως θεσπίζεται ξεκάθαρα ότι όλα αυτά ισχύουν σαν να ήταν όλα αρμοδιότητα της Κομισιόν. Και στο προπολογισμό είναι μάλιστα τμήμα 3 και σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Για τους εκπροσώπους τώρα, ρώτησαν διάφοροι. Εμείς καταφέραμε να περάσει ότι αφενός θα είναι επίτροποι. Δεν θέλαμε τους γενικούς γραμματείς. Τώρα αρμόδιοι από την αρχή είναι οι επίτροποι. Από την άλλη μεριά θέλαμε να έχουμε και εκπροσώπους που θα είναι απληρωτές μάλλον που θα εκπροσωπούν το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θα αποφασίσει τώρα σύμφωνα με το καταστατικό του που για την ώρα είναι η διαδοχική προεδρία. Αυτοί θα δουν ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι. Το έχουμε γράψει έτσι πάντως ώστε μπορούν να είναι και άλλοι εφόσον τους αναθέσει η κυρία Άστον αλλά πρέπει πάντοτε να έχουν κοινοτική νομιμοποίηση μπορεί να είναι το καταστατικό του Συμβουλίου που το επιτρέπει αυτό ή μπορεί να είναι και το άρθρο 33 ώστε να μην είναι ένας υπουργό εξωτερικών ο οποίος να μην έχει επίσημη κοινοτική νομιμοποίηση να μην μπορεί να εμφανίζεται αυτός εδώ ως εκπρόσωπος νομίζω ότι αυτά σωστά τα είπαμε με την γεωγραφική ισορροπία τα είπα Λέει και εδώ ότι η πρόσληψη θα βασίζεται στα προσόντα αλλά και στη βάση μιας γεωγραφικής κατανομής από όλες τις χώρες μέλη και στην επανεξέταση του 2013 θα ληφθούν υπόψη όλα αυτά μαζί με πρόσθετες προτάσεις για πρόσθετα μέτρα για την διόρθωση ενδεχομένων ανισοτήτων παραπάνω πράγματα από αυτά που ε, μέχρι τώρα δέχονταν στο Συμβουλίο οι χώρες οι οποίες είχαν και το δικαίωμα κυρίας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό. Και δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βγάλουμε και παραπάνω. Για την κυρία Λέζινγκ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μυστικές υπηρεσίες ούτε έχει και την πρόθεση, ούτε έχει και την νομική βάση για να δημιουργήσει μυστικές υπηρεσίες. Γι' αυτό νομίζω ότι στερείται η επιχειρηματολογία σας οποιασδήποτε βάσος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τους μεταφραστές που θα φύγουν τώρα. Άρα, Γκουαλτιέρη, αν θέλετε να μιλήσετε, θα πρέπει να μιλήσετε αγγλικά. Yeah, okay. But In English.